So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle. Αγαπητοί συνάδελφοι, hinter uns gebracht. Ένα τρίο τη εργασία το ολοκληρώσαμε μαζί με την Επιτροπή Απασχόληση. Τώρα θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα θέματα. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστώ, ε, να σας ευχηθώ, συγγνώμη, καλή χρονιά. Βεβαίως ε, έχει περάσει ο χρόνος και έχουμε κάνει πολλά πράγματα και έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει πολύ καιρός. Παρόλα αυτά είναι η αρχή ακόμα του χρόνου και θα ήθελα να σας ε, ευχηθώ καλή χρονιά. Χαίρομαι για την συνέχιση της συνεργασίας μας και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει με εξίσου υποκοδομητικό τρόπο όπως και την προηγούμενη χρονιά. Και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν συμπληρώσεις προσθήκες σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Εάν όχι, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται και θα έρθουμε στο σημείο 4 της διάταξη. στην έγκριση των πρακτικών της 9ης Νοεμβρίου, της 23ης και 24ης και 4, Νοεμβρίου και 4ης Δεκεμβρίου, τα πρακτικά της 18ης ε, και 19ης Οκτωβρίου θα τα βρείτε στο φάκελό σας και θα σας πρότεινα τα υπόλοιπα πρακτικά να θεωρηθούν ότι εγκρίνονται. Και τώρα θα έρθουμε στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Υπάρχει διερμηνία σε εξής γλώσσες σήμερα. Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Τσεχικά, Εστονικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Βουλγαρικά και Ρουμανικά. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αποφάσισα το συντονιστών της 4 Δεκεμβρίου ε, σας έχουν αποσταλεί ε, στις 6 Δεκεμβρίου ε, και θεωρούν επισήμως ότι εγκρίνονται εφόσον μέχρι την προθεσμία της 8 Δεκεμβρίου δεν υπήρξαν αντίρρησεις. Και τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρόκειται για το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης και είναι οι προτάσεις μας. Λοιπόν, ε, προτάσεις για μια σύσταση του Συμβουλίου για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για μια υψηλής ποιότητας επαγγελματική κατάρτιση ε, σε σχέση με τη μία πρόταση ψηφίσματος και σύμφωνα με την πρόταση για μία νέα σύσταση Συμβουλίου για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, κατάρτισης, υψηλής ποιότητας κατάρτισης, η Επιτροπή Απασχόλησης αποφάσισε τη, να αποδεχθεί την ε, προθεσμία μας για υποβολή των ε, τροπολογιών ε, αποφασίσαμε να γίνει μέσω ε, επιταχυμένη διαδικασία και η έκθεση αυτή τη στιγμή υπάρχει στα αγγλικά. Το ίδιο ισχύει και για τι ε, τροπολογίε, γιατί ο στόχο τη Επιτροπή Απασχόληση ήταν οι αντίστοιχε συστάσει να υποβληθούν εγκαίρω για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Δηλαδή, η Επιτροπή Απασχόληση θα αποφασίσει τέλη Φεβρουαρίου και εμεί το Μάρτιο στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε για αυτό το σχέδιο ψηφίσματο Γι' αυτό ε, αποφασίσαμε αυτή την ταχεία διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι δικές μας προτάσεις να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή Απασχόλησης. 15 τροπολογίες έχουν υποβληθεί στην ψηφοφορία και αυτό οδήγησε σε 5 συνδυαστικέ ε, τροπολογίες και θα ήθελα σε σχέση με τον κατάλογο ψηφοφορίας θα ήθελα να σας επισημάνω το εξή. Εγώ ως ε, πρόεδρος είμαι σε αυτή, ως σε αυτή τη διαδικασία και σε ορισμένα σημεία θα βρείτε ένα μείον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ με τις τροπολογίες, αλλά πολύ συχνά οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτές τις τροπολογίες ε, αποκλειστικά πρόκειται για καθήλυνα αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης. Και επειδή στις προηγούμενες εβδομάδες ε, ε, διαφωνήσαμε με την Επιτροπή Απασχόλησης ε, για ορισμένα σημεία του κειμένου όσον αφορά κάποιες υπερβάσεις αρμοδιότητας από τη δική τους πλευρά. Εγώ ως πρόεδρος ε, θεώρησα ότι είμαι υποχρεωμένη να τηρήσω αυστηρά τους προβλεπόμενους κανόνες, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από το ίδιο το περιεχόμενο, αλλά ακριβώς από τη τυπική ε, διαδικασία ότι πρόκειται για καθηλυρμοδιότητα της Επιτροπής Άρα όταν ε, δείτε το μείον σε ορισμένα σημεία του κειμένου, σε αυτό οφείλεται. Και πιστεύω ότι μπορούμε άμεσα να περάσουμε στην ε, διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ξεκινάω με την τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε στην τροπολογία επαριθμών 11 με προφορική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία υπαριθμών 14 με, με προφορική, την προφορική τροπολογία 2 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ωραία, θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας ψηφοφορίας. Έξι υπέρ και 16 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία παρθμών 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 με την προφορική τροπολογία παριθμών 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία υπαριθμών 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει υπαλήθευση 31 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. Δεν λειτουργήσε το δικό μου το μηχάνημα, ψηφίζω θετικά. Θα πάω σε άλλο μηχάνημα. Okay. Παρακαλώ βάλτε θετική ψήφο. Yeah. a... Ίσως ε, να πάτε σε άλλο κάθισμα πράγματι also mit 14, 14 zu 10 Stimmen angenommen. 14 προς 10 ε, εγκρίνεται. 35 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Με συγχωρείτε για την 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 35 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 36 έχει αποσυρθεί. Η 37 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 42 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 47 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 με την τροποφορική τροπολογία παρθών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σα ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. δύο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τέσσερα 3 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. πέντε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα θα έρθουμε στην τελική ψηφοφορία η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέραστη ψηφοφορία. 25 ψήφοι υπέρ, μία εποχή εγκρίνεται. Σας ευχαριστούμε και θα, θα διαβιβάσουμε τις τροπολογίες ε, με τη μορφή αυτή στην Επιτροπή Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα έρθουμε στο σημείο της ημερήσιας διάταξης υπαριθμών 7 την έγκριση του ενός σχεδίου γνωμοδότησης για την απαλλαγή στο συνολικό σχέδιο προεπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής και στη συνέχεια την, ε, το σχέδιο ε, για την απαλλαγή 2016 για το μεταφραστικό κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Στροζιεύσκη ήταν ο εισηγητής μας. Θέλετε να έχετε το λόγο. Καλώς τότε θα περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία και θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία υπαριθμών 2. Ε, Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία περιθμών 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία υπερθμών 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Συγγνώμη, το πρώτο τμήμα. Σε τρία τμήματα 21. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Ε, πέρας της ψηφοφορίας, με 24 ψήφους υπέρ και 3 αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Ε, θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Σιγητή. Και τώρα θα πράσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την επόμενη ψηφοφορία που αφορά την ε, απαλλαγή για το κέντρο μετάφρασης. 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και 5. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα πράσουμε στην ε, ηλεκτρονικά στη ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 27 ψήφοι υπέρ, καμία εποχή, καμία αρνητική ψήφο, ομόφωνα εγκρίνεται, θερμά συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Και βεβαίως ε, ε, ευχαριστούμε και τους σκιώδες και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο ημερήσιας διάταξη 9 ε, που αφορά το σχέδιο διαγμα... Ε, γνωμοδότηση για διασυνοριακέ αιτήσει επιστροφή ε, έργων τέχνη και πολιτιστικών αγαθών που λελατήθηκαν σε ένοπλε συγκρούσει και πολέμου. Ε, συνδέομαστε με το άρθρο 54, αρμόδια επί τη ύλη επιτροπή, είναι η νομική επιτροπή. Η συγκριτή μα ο κ. Χουντή. Κύριε Χουντή, θέλετε το λόγο. Όχι. Ωραία, θα περάσουμε άμεσα στη ψηφοφορία. Ένα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Δύο υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά θα ήθελα να το ελέγξουμε πέρας της ψηφοφορίας 14 προς 9 και 4 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθών 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Μπορούμε να το παληθεύσουμε. Ε, συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 προς 9 εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δέκα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. έντεκα, Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμό 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ωραία, να γίνει επαλήθευση για την 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας.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 Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης που αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018. Ε, συντάκτρια είναι η Julie Ward και εδώ συντονιστές αποφασίσαμε μια γνωμοδότηση να στάξουμε μια γνωμοδότηση για την αρμόδια επιστήμη τη Επιτροπή, ε, την Επιτροπή Επασχόληση, και εδώ συμφωνήσαμε να υπάρξει ταχεία διαδικασία, γιατί η έκθεση αυτή θα πρέπει να πάει στην ερηνή συνεδρίαση του Συμβουλίου και εμεί θέλουμε να διεξαχθεί η ψηφοφορία το Μάρτιο. Άρα λοιπόν, τόσο η έκθεση όσο και οι τροπολογίε διατίθενται ε, μόνο στα αγγλικά και η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 26 Ιανουαρίου 10 η ώρα το πρωί. Και βεβαίως ε, οι τροπολογίες στο πλαίσιο αυτής της ταχείας διαδικασίας ε, υπάρχουν μόνο στα αγγλικά. Τζούλι, έχεις το λόγο. Ε, thank you very much, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, η ετήσια έκθεση ανάπτυξης λαμβάνει η χώρα φέτος σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία ε, εγκρίθηκε ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ε, σε ό,τι μας αφορά εμάς εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού η ανακοίνωση του Νοεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ε, εγώ ήμουν υπεύθυνη για την περσινή έκθεση υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια Προσπάθησα εδώ να αποτυπώσω αυτήν τη νέα πολιτική εξέλιξη, η οποία είναι θετική. Η ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη το 2018 δείχνει ότι υπάρχει μια μείωση της ανεργίας, μια μείωση ε, της εγκατάλειψης του σχολείου και τη συμμετοχή στην ανώτερη εκπαίδευση. Αυτά είναι καλά νέα. Όμως ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα ε, και πολύ πιο σύνθετα, διότι αυτή η πρόοδος ε, δεν ήταν προς όφελος ε, με τον ίδιο τρόπο για άτομα διαφορετικών κοινωνικών στρώματων. Οι νέοι άνθρωποι από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν στην ανεργία. Το κοινωνικό τους περιβάλλον επηρεάζει άμεσα και το σχολικό τους περιβάλλον και τις δυνατότητες ε, επαγγελματικής ανέλυξης. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα δεξιοτήτων, ζητήματα προσώπων, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτε ε, ομάδε του πληθυσμού. Αν θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη πολιτική απασχόληση ε, και ένταξη, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα τη εκπαίδευση των ανισοτήτων στην ε, μικρότερη δυνατή ηλικία. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά την ανάπτυξη της απασχόλησης είναι το θέμα τη ποιότητα των θέσεων απασχόλησης. Έχουμε τη νέα ατζέντα για την απασχόληση. Αυτή είναι σημαντική. Θα πρέπει να δοθεί ε, μια μάχη κατά των ε, συμβολέων με μηδενικές ώρες, ε, των εκπαιδεύσεων που είναι εργασία αμυστή ουσιαστικά. Θα πρέπει κάποιες προηγούμενες συστάσεις μας να τις επαναλάβουμε σε ό,τι αφορά τα benchmarks για τη διαβίου μάθηση αλλά και την εφαρμογή μιας εγγύησης για τα παιδιά. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, δεν μπορώ βεβαίως να τα αναφέρω όλα σε αυτή την έκθεση, μιας και υπάρχει και ένα όριο. Ε, υπάρχουν ζητήματα δεξιοτήτων, εκπαίδευση, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και άλλα στοιχεία, τα οποία όμως θα αναδειχθούν στις ε, τροπολογίες. Αναμένω ε, τις συνεισφορές των συνοδέλφων, παρότι είναι σφιχτή διαδικασία, παρότι είναι μόνο στα αγγλικά, ελπίζω να έχουμε πολλές πολλές συνεισφορές από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Τζούλη. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους Σκιώδης για δύο λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Σάντροβα. I would like to Ευχαριστώ να ευχαριστήσω την Τζούλη Βόρτ, την εισηγήτρια, για αυτήν την γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τις συστάσεις της και με αυτά που ανέφερες ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για μια καλύτερη απασχόληση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί και η επικύρωση των δεξιοτήτων ε, και σε ό,τι αφορά τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα το ποσοστό εγκατάλειψης από το σχολείο, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Υπάρχει μια θετική τάση, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη, ε, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, ε, είμαστε πολύ κάτω από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10% δηλαδή. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης στην πρόθεση οριζόντιων δεξιοτήτων, ε, επιχειρηματικότητας, ε, ε κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Υπάρχει ένα σκέλος της ε, γνωμοδότησης που αναφέρεται στην εγγύηση για τα παιδιά. Δεν είναι νέα ιδέα αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε, μάλλον να υλοποιήσουμε τα παρόντα προγράμματα εγγυήσεων, τα οποία έχουν πολλά κενά. Πρέπει ε, να βελτιωθεί η χρήση και τα εργαλεία που υπάρχουν, η χρήση των εργαλείων μάλλον, ε, το Erasmus Plus, ε, τα κοινωνικά προγράμματα. θα υποβάλω λοιπόν σχετικές τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή και εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τζαμπάτσκι. Θέλετε να πάρετε το λόγο, είστε σκιώδης. Όχι. Ωραία. Τότε κυρία Κιμενές. Χιμενές Μπαρμπά. Α, Χιμενές Μπαρμπά. Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Τζούλη για τη δουλειά της. Συμφωνώ μαζί της ε, το ότι να συμπεριλάβουμε τον κοινωνικό πυλώνα ε, κοινωνικών δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί στο εξάμεινο, το ευρωπαϊκό, διότι είχαμε την κρίση, είχαμε αύξηση των ανισοτήτων, αύξηση τη φτώχεια. πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε. Ε, και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό όπλο γι' αυτό, το όπλο τη εκπαίδευση. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να γνωρίζουμε ποιε είναι οι αλλαγέ που έχουν λάβει στις κοινωνίες μας, ε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην παγκοσμιοποίηση, στην ε, τεχνολογική πρόοδο. Θα πρέπει να έχουν νέα όπλα στη διάθεσή τους ε, οι πολίτες για να φτάσουν στην αγορά εργασίας ε, με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θέλουμε μια εκπαίδευση ποιοτική που να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τα ψηφιακά, έτσι ώστε τα παιδιά μας, οι νέοι μας να αντιμετωπίσουν μια αγορά εργασίας η οποία αλλάζει και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και την ανισότητα. Ε, είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δοθούν κίνητρα για την καινοτομία ε, καθώς και για την κινητικότητα μεταξύ των εργαζομένων, να δημιουργούνται έτσι δυναμικές ομάδες εργασίας και κυρίως συμπεριληπτικές ε, αγορές εργασίας. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χιμένες. Κυρία Χουντή, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας και να της δηλώσω την κατανόησή μου διότι επιχειρεί ένα πολύ δύσκολο και τολμώ να πω ακατόρθωτο εγχείρημα. Γιατί ακατόρθωτο. Διότι κατά τα χρόνια που έχει εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει αποδείξει ότι είναι ο πιο αντιδημοκρατικός ευρωπαϊκός μηχανισμός για αντικοινωνικές πολιτικές. Και δεύτερο, ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ο μοχλός αυτός που θα φέρει ανάπτυξη στην Ευρώπη. Προσδοκεί λοιπόν η συγγητριά μας και καλά κάνει και αυτή θα είναι η προσπάθειά μας και τέτοιες τροπολογίες θα καταθέσω αν είναι δυνατόν και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά αν είναι δυνατόν να μπουν ορισμένες επισημάνσεις από τα προβλήματα που έχουμε στο θέμα της παιδείας και του πολιτισμού και σε αυτό τον αόριστο και απροσδιόριστο λεγόμενο κοινωνικό πυλώνα να ενσωματωθούν στην γνωμοδότησή της. Γι' αυτό, αφού είπα ορισμένα πράγματα, για άλλη μια φορά τη συγχαίρω για μια προσπάθεια που ε, ελπίζω να έχει αποτελέσματα, αλλά δεν θα έχει. Δύο κουβεντούλες ακόμα. Και δεν θα έχει, διότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αλλάζει. Έγιναν και άλλες απόπειρες να ενσωματωθούν κοινωνικά θέματα και δεν είχαν επιτυχία. Ας γίνουν τώρα έτσι τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε. Αλλά να έχουμε και συνείδηση ότι δεν αλλάζει. Είπα ότι είναι μηχανισμός που επιβάλλει τις πιο αντικοινωνικές πολιτικές λόγω δημοσιονομικών, δημοσιονομικής πειθαρχία. Τα αποτελέσματα όσο αφορά την ανεργία των νέων, όσο αφορά τα ποσοστά των νέων που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και τα αποτελέσματα εν γέννη από την άποψη ότι σε σχέση με τις δαπάνες για την παιδεία στις μισές χώρες, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχω δει, έχουν δραματικά μειωθεί, το επαναλαμβάνω ίσως, στις μισές χώρες τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δαπάνες για την παιδεία έχουν μειωθεί. Επομένως, η υψηλή δημόσια παιδεία δεν μπορεί να γίνει χωρίς δαπάνες, πολιτισμός με υποχρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει, χρειάζεται διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Θα προσπαθήσω με τις τροπολογίες να στηρίξω αυτά που νομίζω ότι είναι σωστά. Ε, εύχομαι τα καλύτερα. Ε, ευχαριστώ και πάλι την συγγήτρια. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Helga Trüppel. Um, thank you to... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τη Julie Ward υποστηρίζω ακράδαντα την προσέγγιση της. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, και αυτό δεν είναι επιχείρημα κατά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ότι αντιμετωπίζουμε ε, μείωση της ανεργίας και αύξηση της ανώτατης εκπαίδευσης και αυτό θέλουμε να δούμε, αλλά συμφωνώ με την αξιολόγηση σου Τζούλη ότι δεν αρκούν αυτά, διότι λίγο πολύ αυτοί οι οποίοι είναι ήδη ευκατάστατοι, εποφελούνται, αλλά οι μειονεκτικέ ομάδες και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται σε μειονεκτικέ ομάδες και προέρχονται από δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον δυσκολεύονται. Πρέπει να πω λοιπόν σαφέστατα ότι δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση του κυρίου Χουντή, γιατί είναι πάρα πολύ αρνητική. Υπάρχει πρόοδος και πρέπει να δούμε εάν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε την πολιτική πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι το μήνυμά μας και πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς επ' αυτού. Δεν είναι κατά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όλο αυτό. Ε, διαβλέπουμε πρόοδο και ε, ωφέλη, αλλά πρέπει να Είμαστε πολύ περισσότερο κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι, γιατί αυτό είναι το κοινωνικό κοινό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέραν αυτή και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει πρόοδος και υπάρχουν επιτεύγματα. Εάν τα αρνούμαστε και τα μελούμε αυτά, ε, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σωστά συμπεράσματα. Υποστηρίζω λοιπόν ε, τη Τζούλη ακράδαντα, διότι πιστεύω ότι είναι ρεαλιστική και ε, σόφρονη προσέγγιση της και διαπιστώνουμε με την πρόοδο, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε κυρίως το κοινωνικό χάσμα στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εμείς οι πράσινοι είπαμε ήδη ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να επενδύσουμε σε μια κοινή γραμμή, ιδίω στην εκπαίδευση που να σχετίζεται και με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τα προγράμματά μα, το Erasmus Sin, την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αλληλεγγύη. Ελπίζω να την ονομάσουν έτσι. Ε, θα το ψηφίσουμε το Φεβρουάριο. Και φυσικά χρειαζόμαστε και ε, την εγγύηση αυτή. Ε, ε, ευχαριστώ και υποστηρίζω την Τζούλη. Η κυρία Μπίλτ έχει το λόγο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ε. Ναι, με συγχωρείτε. Στην έκθεση αυτή βλέπουμε την αναφορά για τις δεξιότητες των Ευρωπαίων, κάτι που είναι μοναδικό, διότι η γενιά των 20 και 30 ετών είναι αυτή οι οποίοι είναι περισσότερο πτυχιούχοι ε, και ε, έχουν περισσότερο ευέλικτες μορφές εγνασίας. Το παράδειγμα της Ιταλίας είναι πολύ συγκεκριμένο. Ε, αν έχουμε ανεργία πάνω από 30% στην Ιταλία, πώς μπορεί να το θεωρείτε αυτό επιτυχία στους νέους. Ε, φυσικά όλο αυτό υποχρεώνει και τα κράτη-μέλη λόγω των πολιτικών λιτέτατος να μειώσουν τον προϋπολογισμό. Ε, μειώθηκε ο προπολογισμό στην Ιταλία κατά 20% για την εκπαίδευση και κυρίως στο νότο της χώρας ε, τα ποσοστά είναι συγκρίσιμα με τα ποσοστά της Λατινικής Αμερικής στην ανεργία, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι καλό. Οι χώρες του Νότου και η Γαλλία έχουν πέσει στους ε, διεθνείς δείκτες και πρέπει να προσπαθήσουν ε, να προλάβουν αυτές τις καθυστερήσεις. Και εμείς τους ζητάμε να εντάξουν και τις μειονεκτούσες ομάδες, δηλαδή τους μετανάστες. Αυτό φυσικά θα έχει συνέπειες και στα δημόσια οικονομικά και θα μειώσει και το επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη λύση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλες τρεις παρεμβάσεις. Um, Δεν ε, ε, συμφωνώ με την ε, άποψη της εισηγήτριας ότι θέλουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη ταυτόχρονα με την ανάπτυξη στην εκπαίδευση και συμφωνώ μαζί της ότι έχουμε εξάπλωση των ε, συμβολέων επισφαλούς εργασίας, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα. Ε, οι εργοδότες ε, μειώνουν και το κόστος και φυσικά όλα αυτά ε, σημαίνει για τους ανθρώπους ότι το να έχουν κάποια δουλειά είναι καλύτερο από το να μην έχουν καμία δουλειά. Ε, στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες ε, ο αριθμός ρεκόρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν είναι λύση. Στις νότιες χώρες σοβεί η ανεργία, κυρίως των νέων και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερο, να μην ξεκινήσει αυτή ως αγώνας προς το μπάτο. πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υπάρχουν προσλήψεις και ε, να μην ε, δίνουμε αντικίνητρα σε εργοδότες που αλλιώς ε, θα είχαν κίνητρα για να αυξήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους. Η κυρία Λιμπάτσκα για ένα λεπτό. Αυτό είναι γερμανικά, έτσι. Ε, συγχαρητήρια προς την εισηγήτριά μας, την κυρία Ward. Πρόκειται για μια εξαιρετικά προοδευτική γνωμοδότηση και έχετε την πλήρη υποστήριξή μας και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και το γεγονό ότι τοποθετούμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται... υπάρχει εδώ μια πολιτική υποστήριξη. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Δηλαδή, οι χώρες μέλη, ενώ συνεννοήθηκαν για την αύξηση των πόρων, χρειαζόμαστε, λέγοντας ότι χρειαζόμαστε ένα σύμφωνο πολιτισμού, δηλαδή αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση, όχι αμυντικό σύμφωνο. Η Τζούλη τόνισε πολύ σωστά εδώ τη διάσταση αυτή αλλά το να εξετάσουμε το θέμα της εκπαίδευσης μόνο από την ε, προοπτική της αγοράς εργασίας δεν είναι σωστό. Δεν πρόκειται μόνο για τα ποστά απασχόλησης, αλλά και για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Για το γεγονός επίσης ότι θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση να καταναλώνει ε, και ε, να απολαμβάνει τον πολιτισμό. Τώρα, όσον αφορά τις μειονεκτούσες ομάδε, εδώ όντω υπάρχουν πολλά ελλείμματα. Ευχαριστούμε η Σίλβια Κώστα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο κάτι για το συγκεκριμένο θέμα της Ιταλίας. Θα ήθελα να επενθυμίσω στην συνάδελφο Μπίλτ ότι η Ιταλία στα τελευταία τρία χρόνια, χάρη στις κυβερνήσεις κεντροαριστερά, έκανε πολύ περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, στα πανεπιστήμια, υπήρχε και η νομοθεσία για τις θέσεις εργασίας και τα σχολεία από ό,τι με τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις της δεξιάς. Κλείνει η παρένθεσή μου. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Τζούλια Γουόρτ για τη γενεδορία της, για αυτή την επίγουσα διαδικασία και το κείμενό της. Πιστεύω ότι είναι ε, πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ως θετικό το γεγονός ότι το εξάμεινο, και έχει δίκιο ο κύριος Χουντής ότι δεν προσέξαμε στο παρελθόν, αλλά πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει κάτι στην Ευρώπη. Και το είδαμε και με τη συνάντηση ηγετών και στα συμπεράσματα του Γκέτεμπορκ, αλλά και με τη συνάντηση ε, κορυφή στο Δεκέμβριο, που είπαν ότι χωρίς ε, πολιτιστική και εκπαιδευτική πρόοδο δεν υπάρχει πρόοδος και ανάπτυξη. Ε, αυτό για μας ως Επιτροπή Πολιτισμού και ε, πολύ καλά κάνουμε και προσπαθούμε να εντάξουμε τις παρατηρήσεις μας σε συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης και να επαναλάβω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της πρότασης της Τζούλη και μετά θα ε, προτείνουμε και τροπολογίες. Πρώτον, λέει να χρησιμοποιήσουμε τη ρήτρα ευελιξία για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να ε, κάνουν περισσότερε επενδύσει σε παιδεία, σε πολιτισμό και εκπαίδευση. Θεωρώ ότι αυτό είναι ε, καθαρά πολιτικό θέμα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να βγάλουμε από το Σύμφωνο σταθερότητα και τι επενδύσει στον τομέα αυτό. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει διαφορετική προοπτική τώρα και με αυτό τελειώνω γιατί από τις τελευταίες συστάσεις του Συμβουλίου Υπουργών υπάρχουν δύο συστάσεις για τις επενδύσεις για τους διδάσκοντες και ε, να ε, διευρύνουμε σε έναν ευρωπαϊκό τομέα εκπαίδευση για να διευκολύνουμε και μέσω τη ε, ΡΙΚΑΡ και άλλων επενδύσεων τι δυνατότητε για ίσε ευκαιρίε. Διότι ειλικρινά αυξήθηκαν οι ανισότητε το τελευταίο διάστημα και μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω πάλι το λόγο στην Τζούλη. Θέλεις να πάρεις το λόγο. Ε, um, Ευχαριστώ για τα σχόλια, είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Και συμμερίζομαι πολλά από αυτά που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Μικαέλα, αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα πολύ σωστό, αλλά πρέπει να μιλάμε για κοινωνική επιχειρηματικότητα, όχι απλά επιχειρηματικότητα. Είναι σημαντικό αυτό, εάν θέλουμε πραγματικά να συνδέσουμε τους ανθρώπους με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία. Έγινε αναφορά επίσης την κινητικότητα, πολύ σημαντικό και αυτό, το Erasmus και το Erasmus Plus, ε, εδώ παίζουν σημαντικό ρόλο. Επίσης, τα νέα εργαλεία για, τα, για τις νέες δεξιότητες, καινοτομία, σε ένα τοπίο που αλλάζει νέες μορφές εργασίας ουσιαστικά, τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε να φανταστούμε ε, ποιες θα είναι στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να εξοπλίσουμε τους πολίτες με μια σειρά από δεξιότητες οι οποίες να είναι προσαρμόσιμες, να είναι ευέλικτοι στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ευχαριστώ που μας υπενθύμησες ε, το θέμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, πολύ σημαντικό και αυτό και για τη Χέλγα ε, υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα ε, σαφή, δεν, δεν μπορούμε να την ξεχνάμε. Ε, πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι σημειώνεται πρόοδος υπό δύσκολες ε, συνθήκες, αλλά υπάρχει πρόοδος. Βεβαίως ανησυχώ και εγώ για το θέμα της υγείας, της ευημερίας, τις ίσες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους με αναπηρία θα πρέπει να εφαρμόσουμε περισσότερο τα υπάρχοντα μέσα, τα υπάρχοντα εργαλεία που έχουμε στη θέση μας. Είναι σημαντικό εδώ ε, τα κράτη-μέλη να μην αδρανίσουν, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή του. Το καλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι μπορούμε να ανταλλάσσουμε βέλτιστε πρακτικέ. Μπορούμε να μοιραστούμε αυτέ τι καλέ πρακτικέ, να στηρίζουμε οι μεν του δε. Είναι από τα καλά αυτή τη επιτροπή. Άλλωστε, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Μοιραζόμαστε τι γνώσει μα και την πραγματογνωμοσύνη μα. Ε, αναμένω τις τροπολογίες σας και νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία είναι 26 Ιανουαρίου, 10 η ώρα ε, και όπως σας είπα μόνο στα αγγλικά. Καλή επιτυχία όσον αφορά την συνέχιση των εργασιών, αλλά θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, 11 η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας. Και αν είμαι σωστά ενημερωμένη, ήδη έχουν φτάσει οι προσκεκλημένοι μας. Παρακαλώ να έρθουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω θερμά και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά την ε, Βουλγαρική Προεδρία, η οποία εκπροσωπείται από τρεις υπουργούς, δύο υπουργούς και μία, μία υπουργό που είναι αρμόδιοι για τους ε, διάφορους τομείς για τους οποίους είμαστε εμείς υπεύθυνοι εδώ σε αυτή την ε, ε, επιτροπή. Ο κύριος Καζιμίρ Βάλτσεφ, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας στον εκπαιδευτικό τομέα, ο κύριος Κράσεν Κράλεφ, Υπουργός Νεότητας και Αθλητισμού και Υφυπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μέλια Γκρέσεβα ε, τους καλωσορίζω όλους θερμά. Η Βουλγαρική Προεδρία έχει αναλάβει την ε, Προεδρία του Συμβουλίου σε μια δύσκολη εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τόσο εσωτερικά ε, αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις, το Brexit ε, για παράδειγμα, αλλά και στη διεθνή σκηνή βρισκόμαστε ενώπιον σοβαρών ε, προκλήσεων και θα πρέπει να σκεφτούμε για το πώς και με ποιο τρόπο ε, θέλουμε να εξελιχθεί στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκτός τούτου υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα επιτάπητος. Για παράδειγμα, στο δικό μας τομέα, η οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα ε, την οποία ελπίζω θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε εντό τη Βουλγαρικής Προεδρίας. Υπάρχει μια προετοιμασία επίση της συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και εδώ ε, γίνεται μια συζήτηση σε σχέση με το μέλλον των ε, προγραμμάτων για τα οποία είμαστε εμεί αρμόδιοι και έχουμε σημαντικές εκθέσει πρωτοβουλία δρομολογήσει και ε, θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία σειρά λοιπόν σημαντικών ε, θεμάτων. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που η Βολγαρική Προεδρία, η οποία κατέστησε σαφές στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της, ότι πρόκειται να δώσει μεγάλη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης και της ε, κατάρτισης, και θεωρώ ότι αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα και ασφαλώς θα έχει την αμέριστη υποστήριξη ε, της Επιτροπής εδώ. Ε, θα ήθελα να δώσω στον καθένα ε, το λόγο για 10 λεπτά και θα πρότεινα μετά από την κάθε παρουσίαση να κάνουμε, να περιβάλλουμε ένα γύρο ομιλιών για να μην αναμίξουμε όλα τα θέματα στο τέλος. Το κάνουμε λοιπόν σε τρία τμήματα. Θα ξεκινήσουμε για τον Υπουργό Εκπαίδευσης και Επιστήμης, τον κύριο Βάλτσεφ. Καλωσορίσατε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Πέτρα, ουβαζάμι, Δεν... Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και έχω την ε, δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας ε, και να συνεργαστώ για σημαντικά θέματα στον εκπαιδευτικό τομέα. Ε, ασφαλώς υπολογίζω στη δική σας υποστήριξη προκειμένου να έχουμε μια αξιόλογη εκπαίδευση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα για την ε, νεολαία. Ε, το εμβλημά μας είναι ε, ενώση. Γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι μαζί σας θα μπορέσουμε να εργαστούμε για μια ισχυρή Ευρώπη και για την εκπαίδευση πολιτών που θα συμμερίζονται τις αξίες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους από εσά που το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους ε, επισκέφθηκαν πολλές βουλγαρικές πόλεις και ελπίζουμε ότι και τους προσεχείς μήνες θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και άλλα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού. Το έτος 2018 είναι πολύ σημαντικό έτος για τη Βουλγαρία, γιατί η χώρα μας για πρώτη φορά αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία και πρόκειται για ένα έτος κλειδί και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε την πρόταση της Επιτροπής για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο πλαίσιο του Brexit και άλλων σημαντικών προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτό το έτος 2018 είναι έτος κλειδί και για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της ε, εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ε, στο Γκέτεμπορκ ε, υπήρξε μια συνάντηση κορυφής και έγινε και μια συνάντηση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο σε σχέση με τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής. Πριν επισέλθω στις σημαντικές προτεραιότητες ε, της Βουλγαρικής Προεδρίας, επιτρέψατε μου παρακαλώ να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους της Εστονίας γιατί χάρη στην εξαιρετική του συνεργασία η Βουλγαρία μπόρεσε να λάβει την Προεδρία σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο και θα ήθελα να σας ευχαριστώ τόσο και τον κύριο Μαρίνοφ και τον κύριο Μαν για την επιτυχή ολοκλήρωση των ε, ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στις τελευταίες ε, μέρες του 2018 μια συμφωνία για την ψηφιοποίηση και την δημιουργία μια πλαστική πλατφόρμας πολιτών. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, αυστακούς συναδέλφους οι οποίοι έχουν το δύσκολο έργο της ε, του νομοθετικού έργου για το Erasmus Plus καθώς και για τις επικείμενες πρωτοβουλίες της ε, Κομισιόν. Η Βουλγαρική Προεδρία θα στηριχθεί σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες. Δύο εξ αυτών ε, το μέλλον Ευρώπης και οι νέοι, καθώς και η ψηφιακή οικονομία και οι ε, δυνατότητες, οι του μέλλοντος ε, είναι οι πιο σημαντικές. Θα μας απασχολήσει το θέμα των ευρωπαϊκών επενδύσεων στον τομέα της κατάρτισης. Η Βουλγαρική Προεδρία υποστηρίζει την τάση για αύξηση των επενδύσεων και της υπεραξίας του Erasmus Plus προς την κατεύθυνση μιας αύξησης κινητικότητας και καλύτερης ανταλλαγής και καλύτερων πρακτικών μεταξύ μαθητών και διδασκόντων ε, καθώς και την ανάληψη μέτρων για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού νέων ανθρώπων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτισμού για, την, για το φιλόδοξο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους σε σχέση με το μέλλον του προγράμματος. Χαιρετίζουμε την πρότασή σας για μια σημαντική αύξηση του προπολογισμού του προγράμματος, ούτως ώστε το Erasmus ΣΥΝ ε, μέσα τη της ενεργούς των πολιτών, καθώς και την ε, υποστήριξη των ε, ευρωπαϊκών αξιών να μπορέσει να προχωρήσει μαζί με τους συναδέλφους στη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου θα αποφασίσουμε με, ε, για το μέλλον του προγράμματος. Α, θα σε έρθουμε στην διάμεση έκθεση για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ε, θα δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα μια αύξηση της περίληψης των πολιτών και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς την ε, κατάρτιση νέων από νέες περιφέρειες. Είναι σημαντικό να έχουμε μια νέα, ε, νέα στοιχεία για τους πιο ε, χαρισματικούς, πιο ταλεντούχους νέους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, χρειαζόμαστε αντίστοιχα κονδύλια από τον προϋπολογισμό αλλά και τη δημιουργία εταιρικών ε, σχέσεων για την πρόθεση του Εράσμου ΣΥΝ όσον αφορά και τις διαρθρωτικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό τομέα με στόχο μιας υψηλής ε, ποιότητας ε, σχολικό πρόγραμμα. Οι συνέργειες μεταξύ Εράσμου ΣΥΝ και εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών θα οδηγήσουν στην προώθηση διασυνοριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να αφορούν ε, στην, στις ξένες ε, γλώσσες και την ε, εμβάθυνση στις θρησκευτικέ και πολιτιστικές διαφορές στην Ευρώπη και αποφυγή φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων. Ως Προεδρία του Συμβουλίου έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να διανοιχθούν νέα θέματα, όπως για παράδειγμα αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων. Τα επόμενα βήματα θα γίνουν στη δεύτερη συνάντηση υπουργών στις 15 Φεβρουαρίου. Με χαρά μου διαπιστώνω ότι το Κοινοβούλιο μέσα της Κυρίας Λιμπάτσκα πήρε θέση των θεμάτων αυτών έμφαση δόθηκε στην ανάληψη καταλήλων μέτρων ε, στον τομέα της ψηφιοποίησης, της ε, γνώσης για τα μέσα και την ε, επαρκή νομοθεσία για την τεχνητή νομοθεσία, ε, για την τεχνική συγγνώμη, νοημοσύνη. Κατά τη διάρκεια της Βολγαρικής Προεδρίας θα στηριχθούμε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Κατάρτιση. ψηφιακές τεχνολογίες προποθετούν κάποια περαιτέρω βήματα όσον αφορά και την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διδάσκοντε θα πρέπει να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, αλλά δυστυχώς στην πράξη πολλές φορές οι νέοι διδασκόμενοι είναι πολύ πιο προχωρημένοι στον τομέα αυτό από τους διδάσκοντες. Χρειαζόμαστε λοιπόν την αύξηση των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο του fake news, για παράδειγμα. Τέλο μέσω τη ψηφιοποίηση δημιουργείται μια ε, κοινωνική ε, ανισότητα, η οποία αντιθέτω θα πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσει για γυναίκες, για παράδειγμα. Οι ψηφιακέ δεξιότητε είναι το θέμα ε, ενό σημαντικού συμποσίου ε, Educated to Create για, την ψηφια... για τις ψηφιακές ε, χρήσεις. Οι ψηφιακές ε, γνώσεις είναι μία από τις αρμοδιότητες κλειδί το Φεβρουάριο θα ξεκινήσουμε με την ε, προσαρμογή του πλαισίου που υπάρχει από το 2006 με συμπερίληψη των νέων τεχνικών και κοινωνικών συνθήκων. Η σύσταση θα συμπεριλάβει κάποιες αλλαγές όσον αφορά την πολυγλωσία, την πολυπολιτισμικότητα, ε, και το πλαίσιο αναφοράς για ψηφιακές ε, δεξιότητες. Ε, και καινοφανές στοιχείο θα είναι όχι μόνο ότι θα ορίζονται οι αρμοδιότητες, οι βασικές αρμοδιότητες, οι αρμοδιότητες κλειδί ε, στη σύσταση αυτή, αλλά και οι καλύτερες πρακτικές για τη χρήση αυτού του, για την αξιοποίηση αυτού του πλαισίου από τις χώρες ε, μέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης για τον κάθε πολίτη και για την κάθε ηλικιακή ομάδα. Όταν μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εστιάζει μόνο στην εσωτερική αγορά, αλλά στηρίζεται και σε κοινέ αξίες. Οι κοινέ αξίες ε, εδραιώνονται στο άρθρο 2 ε, των συνθηκών και είναι ε, ε, καθοριστικές ε, τόσο για μας όσο και τις μελλοντικές γενιές. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα ούτως ώστε να διατηρηθούν στις μελλοντικές γενιές ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινή κληρονομιάς του στην ΑΕΗ να γίνουν ενεργοί πολίτες μιας νέας Ευρώπης. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Έτσι, οι χώρες μέλη θα ενισχυθούν στις προσπάθειές τους για την δημιουργία κοινωνιών συνοχής, την πρόθεση της εκπαίδευσης με συμπερίληψη όλων των πολιτών και αποφυγή φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης. Η ευρωπαϊκή κοινωνία εξελίσσεται ε, στο πλαίσιο μιας όλο και μεγαλύτερης ε, πολυπολιτισμικότητας και ε, πολυγλωσίας. Θα πρέπει να εμπνεύσουμε περισσότερους πολίτες, πιστεύουμε, για το επάγγελμα του διδάσκοντος. Η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχει ένα μηχανισμό για τη διοργανική συνεργασία όσον αφορά την ε, ε, εκπαίδευση. Για μας ε, είναι σημαντικό να ελέγχουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών οι οποίοι ταξιδεύουν και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να έχουν και μια, τη δυνατότητα μιας ε, συνεχούς ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όλα αυτά τα θέματα είναι καθοριστικά για το όραμα της ε, Ευρώπης στο εγγύς μέλλον. Γι' αυτό υποστήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να υπάρξει μια συνένεση ε, έχει ένα ρόλο κλειδί στο πλαίσιο της Βουλγαρικής ε, Προεδρίας η οποία θα μεριμνήσει για σημαντικές διοργανώσεις στη Βουλγαρία στον τομέα της εκπαίδευσης και θα χαρώ για την συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάλτσεφ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και περιεκτικό πρόγραμμα για τους προσεχείς έξι μήνες και νομίζω ότι πολλά από τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε συμφωνούν και με τις δικές μας ε, προτεραιότητες που έχουμε εδώ στην Επιτροπή. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχήν στους συντονιστές για τρία λεπτά το πολύ και στη συνέχεια θα έχουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων και εάν ε, τα ανάγκη μια δεύτερο, ένα δεύτερο γύρο. Κύριε Σαμπίνε Φερχάν, ε, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που ε, ε, εγκρίνατε και τις δικές μας ε, προτάσεις ή μάλλον είστε ευνοϊκοί απέναντι στις δικές μας προτάσεις ε, προσεχώς η Κομισιόν θα συζητήσει το μέλλον του προγράμματος Erasmus Plus και εδώ μια, προβλέπεται μια αύξηση των πόρων. Ε, έχουμε ποστά αποτυχίες 18-20% των, μόνο 18-20% των προγραμμάτων που μπορεί, μπορούν να εγκριθούν την χάνουν χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ ένα σημαντικό έλλειμμα της χρηματοδότησης. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να πολλαπλασιάσετε εδώ τον προπολογισμό, να ενισχύσετε τον προπολογισμό, γιατί τα μέσα είναι πενιχρά. Ε, αυτή τη στιγμή ε, κυριαρχεί το ζήτημα στο Εράσμος της ανταλλαγής φοιτητών, εγώ θα ήθελα εδώ να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης, vocational training, ούτε ώστε να έχουμε εγκαίρως μια ανταλλαγή μεταξύ μαθητών για να προετοιμάσουμε και τους ε, μαθητές. Επίσης και ανταλλαγή ε, των καθηγητών, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να εξοικειωθεί με τις best practices, τις βέλτιστες πρακτικές και για τους ε, καθηγητές. Και να υπάρξουν, ε, υπάρχει εδώ μια ενίσχυση των προγραμμάτων γιατί θεωρώ ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αποδοχή των προγραμμάτων. Ίσως θα μπορούσατε να σχολιάσετε εδώ γιατί η Βουλγαρική Προεδρία ε, βεβαίως ε, μέσω της, ε, του Συμβουλίου συμμετέχει στον προγραμματισμό. Ευχαριστώ, Σίλβια Κώστα. Καταρχάς, να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για αυτή την πρώτη Προεδρία που είναι ιστορική στιγμή για την χώρα σας και ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Το 2018 είναι έτος κλειδί και είναι έτος κλειδί, θα το πούμε και αργότερα, γιατί είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που συνδύει δέει όλο και περισσότερο ε, εκπαίδευση και πολιτισμό. Θα συμμετέχει η Προεδρία σας ε, όλο και περισσότερο στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που αφορούν το Erasmus ΣΥΝ. Ξέρετε ότι έχουμε εκφράσει την άποψή μας και ζητάμε πολλαπλασιασμό των πόρων και η ομάδα μας ε, ε, συμμετείχε στην εκστρατεία 10 φορές Εράσμους, 10 times Εράσμους, διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια φιλοδοξία για να προσεγγίσουμε όλο ένα και περισσότερους νέους και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γραμμές του προγράμματος να περιλαμβάνουν και ε, ε, μέσα ένταξες. Εμεί προτείναμε την ιδέα του ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής ε, Φοιτητική κάρτας που θα έχει μεγαλύτερη πρόσβαση, αλλά θέλουμε να εντάξουμε και άτομα με αναπηρία, νέους μετανάστες, ε, αυτά ε, συμπεριλήφθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια και στο πρόγραμμα Εράσμους. αναφέρομαι και στο θέμα της προσβασιμότητας και τη δυνατότητα των σχολείων και των διδασκόντων και ε, το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρό στοιχείο νεότητα στο πρόγραμμα. Μετά από τη Σύνοδο Κορυφή του Γκέτιμπορκ, ε, τι δύο συστάσει που αναφέρατε εσεί του Συμβουλίου, που ελπίζω να εγκριθούν ε, στη διάρκεια τη Βουλγαρική Προεδρία, ε, υπάρχει ε, επιτέλου η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση που δεν υπήρχε στην αρχή αυτή τη θητεία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένε φορέ και όχι επαρκώ από πλευρά Συμβουλίου ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμό είναι θεμελιώδει πτυχέ ε, του, του κοινωνικού θεματολογίου αλλά και τη κοινωνική καινοτομία. Πρέπει λοιπόν να δούμε και το θέμα των πολιετών προγραμμάτων ξεκινώντα από αυτή τη συνειδητοποίηση και πρέπει να είναι οριζόντιο αυτό σε όλε τι πολιτικέ. Το άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι το θέμα της δυνατότητας να υπάρχει ένα πραγματικό σχέδιο δράση, το οποίο προβλέπεται όσον αφορά τι ψηφιακέ δεξιότητε, γνωρίζοντα όμω ότι πρόκειται και για δεξιότητε υψηλού επίπεδου, όχι μόνο ε, τι άμεσε δεξιότητε που χρειάζονται για την ε, αγορά εργασία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι και σε 10 χρόνια τα παιδιά τα οποία θα εγγραφούν τώρα στο σχολείο θα ε, κάνουν τα μισά από τα μαθήματά τους με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ε, και είδα και στο πρόγραμμά σας, ε, και με αυτό ολοκληρώνω, θέλετε να υποστηρίξετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για μεγαλύτερη σύμπραξη μεταξύ πανεπιστημίων, ώστε ευθύς εξ αρχές να έχουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, ε, κοινά πτυχία δηλαδή και κοινά προγράμματα σπουδών, ίσως και σε δύο γλώσσες. Αυτό για μας είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Τζαμπάτσκι. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω. Ε, ε, έχετε ένα δύσκολο έργο μπροστά σας. Το γεγονός ότι μπορείτε να μιλήσετε τη μητρική σας γλώσσα στην αίθουσα αυτή είναι κάτι αξιοσημείωτο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία κύριε και, κύριε θα ήθελα να απευθύνω το εξή ερώτημα προ εσά σε σχέση με τι νέε τεχνολογίε στον τομέα τη εκπαίδευση και όσον αφορά τη δική σα θέση εδώ. Αναμφίβολα, οι νέε τεχνολογίε θα πρέπει να προωθηθούν στον τομέα τη εκπαίδευση και όχι να αποφευθούν. πόσο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τους καθηγητές για τη χρήση νέων τεχνολογιών ε, είπατε είναι σημαντική προτεραιότητα γιατί οι καθηγητές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους μαθητές όσον αφορά τις ικανότητες. Όσον ε, τι πιστεύετε για την εισαγωγή ηλεκτρονικών διδακτικών εγχειριδίων, διδακτικών βιβλίων. γιατί πιστεύω ότι αυτό θα διευκόλυνε την κινητικότητα ε, γιατί ε, με τον τρόπο αυτό λύνονται και κάποια θέματα αλφαβήτου, όπως είναι το κυριλικό αλφαβήτο, το δικό μας. Τι λέτε για τις ε, συμφωνίες όσον αφορά την ε, αναγνώριση των ε, γλωσσών ε, στα οποία αποκτώνται τα διπλώματα στην Ευρώπη. Η Χέλγα Τρούπελ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τη Βουλγαρική Προεδρία που μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Η πρώτη μου ερώτηση δεδομένου ότι είμαι και σκιώδης για τους πρασίνους, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι ε, κατά πόσον η Βουλγαρική Προεδρία ως Προεδρία θα υποστηρίξει τη θέση του Κοινοβουλίου των ε, δύο εισηγητών, Όλμπρικτ από το ΕΛ και Τούμα, το Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ε, για προπολογισμό με αύξηση κατά 3%. Εσείς υποστηρίζετε τα αιτήματά μας ως Επιτροπή Πολιτισμού να αυξήσουμε τα κονδύλια για το Εράσμου ΣΥΝ, τον πολιτισμό, την Ευρέπη για τους πολίτες και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα λέγεται έτσι. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να λέγεται Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αλληλεγγύης. Θα ε, κάνετε αύξηση στον προπολογισμό για να είναι επιτυχή αυτά τα προγράμματα στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, επειδή το θέμα μας είναι παιδεία και είμαστε στη διαδικασία ε, οριστικοποίησης της μεταρρύθμισης για τα πνευματικά δικαιώματα, το ερώτημα λοιπόν είναι αν οι Ευρωπαίοι πολίτες και κυρίως οι νέοι θα αναγνωρίσουν ότι ε, δεν μπορούμε να έχουμε ε, δημοσιογραφία ποιότητας ε, και πολιτιστική ποικιλομορφία ε, χωρίς αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πληρώνεται το περιεχόμενο. Το γεγονός δηλαδή ότι ο κόσμος θα πρέπει να πληρώνει αν θέλουν να απολαμβάνουν ποιοτική δημοσιογραφία και ποικιλομορφία. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλο. Όχι, κυρία Μπίλτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Μιλάμε πολύ για την κινητικότητα. Το θέμα με την κινητικότητα είναι όμως και η διαρροή ε, εγκεφάλων. Χιλιάδες ε, Βούλγαροι ε, εξαιρετικά καταρτισμένοι φεύγουν από τη χώρα προς άλλες χώρες της Ένωσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσες δεξιότητες και φεύγουν από τη χώρα, πώς καλύπτεται αυτό το κενό. Θα ενισχύσετε τις ε, οι προϋποθέσεις ε, εισόδου στο Εράσμους ε, και θα επανεξετάσει την πολιτική για την μπλε κάρτα και ποιες θα είναι οι νέες προϋποθέσεις. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, για λόγους πολιτικής αυρότητας οφείλω να ευχηθώ στον Βούλγαρο Υπουργό και γενικώ στη Βουλγαρία να έχει μια πετυχημένη Προεδρία και τον ευχαριστώ για τις παρουσίαση των προτεραιοτήτων στον τομέα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Είμαι από την Ελλάδα, αν, για να έτσι λίγο να γνωριστούμε καλύτερα. Ε, θέλω να πω ότι ε, παρατήρησα ότι στην εισαγωγή <clears throat> επικαλέστηκε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ελεύθερη αγορά, αλλά είναι και αξίες. Και μάλιστα επικαλέστηκε και τα άρθρα του, των συνθήκων η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι αξίες έχουν πάει περίπατο. Ιδιαίτερα αυτές τις οποίες θα επικαλεστεί προφανώς το έργο του ε, ε, η Ευρωπαϊκή Προεδρία, η Βουλγάρικη Προεδρία και είπα ότι είμαι από την Ελλάδα, η αξία της αλληλεγγύης έχει πάει περίπατο. Είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις όλο και περισσότερο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλώ όχι μόνο για την οικονομία. Αλλά για να είμαι μέσα στο θέμα, ε, το κεντρικό πρόβλημα κύριε Υπουργέ, όπως καταλάβατε, ή κατά τη γνώμη μου στο θέμα αυτό είναι το θέμα της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων ε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω τελειώνοντας αυτή την παρατήρηση, επαναλαμβάνοντας τις ευχές να κάνετε ό,τι μπορείτε, στη χώρα σας πόσο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης και δεύτερο, ποιος είναι ο αριθμός των νέων επιστημόνων που φεύγουν από τη Βουλγαρία γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κεντρικά θέματα και γι' αυτό σας ρωτώ τι γίνεται και στη δική σας τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνω το πρώτο γύρο και θα έχουμε στη συνέχεια ένα δεύτερο γύρο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Υπουργέ να προσπαθήσετε σε 4-5 λεπτά να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, σας είπα, ένα σημαντικό στόχος της Βουλγαρικής Προεδρίας είναι η αύξηση των επενδύσεων και εξασφάλιση μιας καλύτερης ε, πρόσβασης στο Εράσμος. Όσον αφορά το ερώτημά σας, για την ε, αύξηση των χρηματοδότησης. Αυτή ήταν και μια ερώτηση της κυρίας Τρούπελ άλλωστε. Θα ήθελα να πω το εξή. Θα αυξήσουμε τις επενδύσεις, δηλαδή θα ενισχύσουμε ε, το αίτημα αυτό στο Συμβούλιο, συνάντηση του Συμβουλίου και θα το συζητήσουμε με τους Υπουργούς ε, Οικονομικών. Και βεβαίως επίκενται διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι υπουργοί μας ε, οικονομικών θα πρέπει να λάβουν σημαντικές απόψεις και σε άλλους τομείς, αλλά θα προωθηθεί ε, το ζήτημα αυτό, η εκπαίδευση δηλαδή. Όσον αφορά τη συμμετοχή διαφόρων ομάδων νέων ή κατηγοριών ε, νέων, σε σχέση με το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης για τους μετανάστες, το οποίο ανέφερε η κυρία Κώστα, και για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Και για τις ομάδες αυτές βεβαίως είναι αναγκαίο να ληφθούν ε, μέτρα. Σημαντική θα είναι και η συμμετοχή των ε, καθηγητών, των διδασκόντων στο πρόγραμμα αυτό. Και βεβαίως θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, ψηφιακή ατζέντα Όσον αφορά τον κύριο Τζαμπάσκι και τις ερωτήσεις για τις νέες τεχνολογίες, θεωρούμε ότι είναι παρέγκλητες και θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να ενισχύει και η χρήση τους από τους διδάσκοντες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ε, προγράμματα για την ενεργοποίηση των καθηγητών, ε, για την χρήση νέων ε, ψηφιακών τεχνολογιών. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί, δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε εντελώς την βιωματική μάθηση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική πρόσβαση στα διδακτικά εγχειρίδια υπάρχουν ήδη στην ε, Βουλγαρία, έχουν επιπρόσθετα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τις δυνατότητες ηλεκτρονικής πρόσβασης ε, ε, στα διδακτικά βιβλία Επίσης υπάρχει μια πολιτική για την εκμάθηση της βουλγαρικής ε, γλώσσας ε, σε άλλες, ε, γλώσ... χώρες. Τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν ληφθεί κάποια επιπλέον μέτρα στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και ιδρύσαμε ένα κέντρο για την ηλεκτρονική εκπαίδευση ή εκπαίδευση εξ αποστάσεως στη Βουλγαρία προκειμένου, ε, και δώσαμε τη δυνατότητα στα σχολεία στο εξωτερικό να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα αυτής της εξαποστάσεως εκπαίδευσης με σκοπό την ε, ε, προσήλκυση των νέων στο χώρο αυτό. Ε, έχω υποστηρίξει το αίτημα για την ε, ε, συμπερίληψη των βουλγαρικών σαν μια γλώσσα για το απολυτήριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Χουντή για το ερώτημά του. Έχουμε έναν ενδιάμεσο προπολογισμό για εκπαιδευτικούς στόχους. Οι δαπάνες εδώ θα αυξηθούν και οι αποδοχές των του παιδαγωγικού προσωπικού θα διπλασιαστούν. Το, η πιο σημαντική πρόκληση ήταν να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση, κυρίως τη μετανάστευση, την έξοδο των νέων ε, τα τελευταία χρόνια από τη Βουλγαρία. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, σημειώνεται μία μείωση αυτών των ποσοστών και με την αύξηση της ε, σύγκλησης τους ε, ε, λόγω τομής έχουμε μια καθαρή μετανάστευση με πρόσημο αρνητικό. Δηλαδή πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι ξεχάσατε την ερώτηση της κυρίας Τρούπελ για το copy word για το copyright. Δεν ξέρω αν είστε εσύ αρμόδιος ή συνάδελφοί σας. Ωραία, θα κρατήσουμε την ερώτηση αυτή και θα επανέλθουμε. Και τώρα θα έρθουμε στο δεύτερο γύρο και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκοφ. Παρακαλώ να περιοριστείτε εδώ στο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κυρία Υφυπουργέ, ε, καλή επιτυχία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Πώς έχει προχωρήσει η Βουλγαρία στην επεξεργασία ενός συστήματος για την ε, τυποποίηση των ε, γνώσεων στην θελοντική εργασία. Ίσως ε, μελλοντικά το σύστημα αυτό της αναγνώρισης θα είναι πολύ καθοριστικό για την επιτυχία του προγράμματος για τις δεξιότητες. Πώς έχει προχωρήσει η Βουλγαρία στον αφορά την εκπόνηση μιας διεθνούς στρατηγικής για την προώθηση ψηφιακών γνώσεων γιατί αυτό έπρεπε να γίνει το περασμένο έτος γιατί ε, μέχρι στιγμής μόνο ένα μικρό ποσοστό των θέσεων εργασίας προποθέτουν ε, ε, ψηφιακές δεξιότητες. Αν επενδύσουμε εδώ στις ψηφιακές δυνατότητες θα βελτιωθούν και οι οι επαγγελματικές ευκαιρίες των νέων. To, to the other ministers, we make it later. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. κύριε. Thank Thank you you very much. Uh, Sorry. very much. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το θέμα της νεολαίας και των μέλλον της Ευρώπης ε, είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της Βουλγαρικής Προεδρίας και όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι στα χέρια των νέων μας και εκεί πρέπει να επενδύσουμε, να επενδύσουμε στο μέλλον τους και να επενδύσουμε βεβαίως και σε μια ποιοτική εκπαίδευση. Χαίρομαι που ακούω ότι συμφωνούμε ε, στο γεγονός ότι οι καθηγητές είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ε, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Πρέπει να τους ε, ενισχύσουμε, πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο τους. Επίσης θα πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές. Στην υποδομή της εκπαίδευσης έχω δύο ερωτήσεις πώς η Βουλγαρική Προεδρία ε, θα μπορέσει να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να επενδύσουν περισσότερα στην εκπαίδευση και το δεύτερο ε, έχει να κάνει με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξέρετε, ολοκληρώνεται φέτος η στρατηγική EU. Τι θα γίνει μετά το 2018 σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Νέους. Τι προτείνετε εσείς. Watts. Η Julie Watts έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα απλώ να αναφερθώ στο θέμα της επιστήμης και να κάνω ένα αίτημα σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται βελτίωση της ε, εκπαίδευσης ε, ε, σε ό,τι αφορά την επιστημονική εκπαίδευση και να συμπεριληφθούν βεβαίως και περισσότερες γυναίκες στη διαδικασία να μην ξεχνάμε και τις τέχνες. Είναι σημαντικό να έχουν ολοκληρωμένη παιδεία οι νέοι. Ε, η επιστήμη ε, χωρίς ε, δημιουργικότητα, χωρίς καινοτομία, χωρίς φαντασία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι δημιουργικοί οι επιστήμονες εξορισμού, διότι πρέπει να σκέφτονται πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, πρέπει να σκεφτούν διαφορετικά. Ξέρουμε ότι επίσης πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους η μουσική, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούν αριθμούς. Ε, οι σχεδιαστές. Ε, υπάρχει λοιπόν ένας διαχωρισμός, ο οποίος είναι τεχνητός μεταξύ των μαθημάτων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δώσει έμφαση και στο θέμα των τεχνών. Κριστίνα Λιμπάτσκα έχει το λόγο τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Προ... ε, Υπουργέ, θα ήθελα να συγχαρώ. Σας άκουσα με μεγάλη μου χαρά. Έχω δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι προτείνεται μια ε, ταχεία εκπαιδευτική διαδικασία για τους ε, πιο νέους, πιο μαθητές. Δεύτερον, η Κομισιόν πρότεινε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα επιστημονικά μαθήματα. Ευχαριστώ θα μετατοπίσω στη συζήτηση σε μια πτυχή που δεν συζητήθηκε. Το Δεκέμβριο του 2016 το Κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής μας με μεγάλη πλειοψηφία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα ε, πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής ε, ε, συνεκτικό για την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία που να έχει μια σαφή σύνδεση μεταξύ στρατηγικών στόχων και γενικών προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Βουλγαρική Προεδρία στα πλαίσια των προτεραιοτήτων τη σκοπεύει να υποστηρίξει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία έχουν διτή αξία, αλλά έχουν και καθήκον να συμβάλλουν στην οικονομία τη Ένωση, όσον αφορά την απασχόληση, τι επενδύσει, την ανάπτυξη και την καινοτομία και επομένως να είναι ε, αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω. Υπάρχει για παράδειγμα το νέο ε, πλαίσιο εργασίας ε, ε, τεσσάρων ετών για το 2019-2022 και τέλος ε, υπάρχει και το θέμα για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το ρώτησε η κυρία Τρούπελ. Υπάρχουν αντίστοιχα των διπλωμάτων ευρασιτεχνίας για την τεχνολογία, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή η Βουλγαρική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ έχω την εντύπωση Έχω όμως την εντύπωση ότι αυτή είναι μια ερώτηση η οποία απευθύνεται στην ε, Υφυπουργό κυρία Γκέσεβα. Θα τη φυλάξουμε. Ο κύριος Σάντεμαφ. Ένα λεπτό. Ε, αξιότιμα κύριε Υπουργέ, καλωσορίστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Βάλτσεφ, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των μαθητών, των πολιτών, είναι μια προϋπόθεση της ανάπτυξης μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας. Δύο ερωτήματα. Τι μέτρα θα προτείνατε για την υποχρεωτική εκπαίδευση και για την μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου. Δεύτερον, η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται άμεσα από την ε, επαρκή επαγγελματική προετοιμασία των καθηγητών και από τις ικανότητές τους. Οι καθηγητές θα πρέπει να χαίρουν με καλύτερης κοινωνικής υπόλοιψης, ούτως ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους τι θα προτείνατε για να αυξήσετε τις ε, επαγγελματικές ικανότητες των διδασκόντων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία... Τα, Θα πρέπει να δούμε ε, πώς ε, θα τα καταφέρουμε με το χρόνο μας, γιατί είναι, υπάρχει μια πληθώρα σημαντικών θεμάτων εδώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γερνέκοφ για το ερώτημά του και για την ε, ε, προώθηση της, ε, των ψηφιακών δεξιοτήτων ως συνώνυμη με την ανάπτυξη ενός ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως είπε. Χρειαζόμαστε βεβαίως μια γενιά η οποία δεν θα είναι μόνο ψηφιακοί χρήστες, αλλά και ψηφιακή δημιουργή. Και σε εθνικό επίπεδο έχουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για ε, ε, ε, όσον αφορά την πληροφορική που συμπεριλαμβάνει μαθητές και με τον τρόπο αυτό θέλουμε να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες ε, στους μαθητές. Όσον αφορά τον κύριο Μπόσκοφ και τις ερωτήσεις του, θα ήθελα να πω το εξή. Θα δράξω την ευκαιρία να σας καλέσω αύριο σε μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τους ε, καθηγητές. Οι επενδύσεις στο διδακτικό προσωπικό είναι σημαντική προϋπόθεση για την βελτίωση των εκπαιδευτικών ε, αποτελεσμάτων στο μέλλον. Και εδώ θα περάσω στο ερώτημα του κυρίου Αντέμοφ, το δεύτερο ερώτημά του. Είπε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στις επικοινωνίες και κυρίως να ενεργοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους, να τους παράσουμε τα κίνητρα, ούτως ώστε να στραφούν προς το επάγγελμα του καθηγητού, του διδάσκοντος. Αυτός είναι σημαντικός ε, στόχος για μας. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε για υψηλή ποιότητα παιδαγωγικό προσωπικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Λιπάτσκα. Η συζήτηση αυτή μένει ανοιχτή. Θα την διεξάγουμε με τους συναδέλφους υπουργούς το Φεβρουάριο. Όσον αφορά και την κυρία Watts, θα ήθελα να πω ότι είναι αναμφίβολο ότι η εκπαίδευση στον επιστημονικό τομέα θα πρέπει να βελτιωθεί. Και ε, το ζήτημα της δημιουργικότητας αυτό αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων κλειδί, ενίσχυση και των ε, παραδοσιακών μαθημάτων, αλλά και εξωσχολικές δεξιότητες. Είχα μια συζήτηση σε σχέση με, τα, με το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε εξωσχολικά μέτρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την ε, ανάπτυξη της ε, επιστήμης στον ευρωπαϊκό χώρο και τη συμπερίληψή της στην εκπαίδευση. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα του κυρίου Αντέμοφ, τα μέτρα δηλαδή για την ε, μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου, εδώ θεωρούμε ότι είναι βασικός στόχος των ε, σχολείων η αποφυγή αυτού του φαινομένου. Το κράτος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε το μηχανισμό για μία προβλέψει τον μηχανισμό για μια ε, συνεργασία των θεσμικών οργάνων, ούτω ώστε να μειωθούν τα ποσοστά εγκατάλειψη του σχολείου. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα πολιτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα προκειμένου να υποστηρίξουμε τα παιδιά αυτά. Ελπίζω να απάντησα όλε τι ερωτήσει που μου θέσατε και θα ήθελα να με συγχωρέσετε εάν παράληψα κάποια ερώτηση. Ναι, α, την ερώτηση του κυρίου Μοργκάνο. Όπως αναφέρθηκε ήδη, το είπα και στην κυρία Τρούπελ άλλωστε, αναμένουμε την πρόταση της Επιτροπής για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο το μήνα Μάιο. όπου θα καταλήξουμε στα πρώτα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Βάλτσεφ, που ήρθατε εδώ, που μας παρουσιάσατε τις ε, προτεραιότητες στον τομέα επιστήμη και εκπαίδευση και έχουμε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή μας. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ίσως θα έπρεπε να κάνουν τις παρουσιάσεις τους πρώτα και οι τρεις υπουργοί και μετά να ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Ε, νομίζω ότι αυτό, γιατί αλλιώς θα, ε, ε, ενδεχομένως θα περικοπεί ο χρόνος της τελευταίας ε, παρουσίας της κυρίας Υφυπουργού. Άρα λοιπόν να ακούσουμε τις δύο παρουσιάσεις τη μία μετά την άλλη και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο γύρος των ερωτήσεων και προς τους δύο υπουργούς. Ο κύριος ε, Κράλεφ, Υπουργός ε, Νεότητας και Αθλητισμού. Θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ. Κύριε Κράλεφ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια τιμή για μένα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας στον τομέα αθλητισμού και νεότητας κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας έχει τεράστια σημασία για μας να έχουμε ένα αποτελεσματικό και διαρθρωμένο διάλογο με το Κοινοβούλιο που συνομοθετεί. Το μέλλον της, των νέων της Ευρώπης συμπεριλαμβάνεται στις βασικές προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Εκτιμούμε πάρα πολύ, θα εκτιμήσουμε μια συνεχή επαφή με εσά με στόχο να καταλήξουμε σε ε, ε, στην επίτευξη το στόχο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις προτεραιότητες μας εδώ, θέσαμε την έμφαση στην ανάπτυξη της ε, πολιτικής για τους νέους. Ε, παρακολουθούμε την εξέλιξη της νεολαίας και έχουμε συνείδηση των ε, προκλήσεων στο χώρο αυτό. Υπάρχουν ταχύες εξελίξεις στις τοπικές κοινωνίες. Η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση, τα μεταναστευτικά ρεύματα, τα φαινόμενα τρομοκρατίας, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας θέτουν τις κοινωνίες μας σε πίεση, οδηγούν σε φαινόμενα επιθετικότητας και ριζοσπαστικοποίηση μεταξύ των νέων το ε, προσπαθούμε να κατατείνουμε προς την οικοδόμηση μιας ασφαλούς και ειρηνικής κοινωνίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε θετικές προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για να συμβάλλουν στην ε, επίτευξη συνοχής και ειρήνευσης στην κοινωνία. Η Βουλγαρία γνωρίζει τις δημογραφικές, δημογραφικές τάσεις μεταξύ της νεολαίας. Γι' αυτό δίνουμε έμφαση στην προώθηση του δυναμικού της νεολαίας και, των ταλέντων της, ούτε ώστε να μπορέσει η δημογραφική τάση να αποκτήσει θετικό πρόσημο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε νέους ανθρώπους γιατί είναι τα προπόθεση ε, θεμολίωσης ενός ε, βιώσιμου μέλλοντος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στον τομέα της εκπαίδευσης των σχολείων και της απασχόλησης ε, για νέου ανθρώπου να γίνουν σημαντικέ επενδύσει. Η Βουλγαρική Προεδρία θέλει να αυξήσει τη συνείδηση για τι δημογραφικέ αλλαγέ εντό τη Ευρώπη. Τα, γιατί θα πρόκειται να επηρεάσουν όλο και περισσότερο τα κοινωνικά συστήματα, ιδιαίτερα τους νέους. Θα συμβάλλουμε ενεργά στην εφαρμογή πρωτοβουλίες για έναν διαφορεμένο διάλογο ως αποτελεσματικό εργαλείο συμμετοχής των νέων ε, και ή δυνατόν έχουμε άμεσο διάλογο μεταξύ νέων ανθρώπων και φορέων λήψη αποφάσεων ε, για παροχή πληροφοριών σε σχέση με την πραγματική κατάσταση νεολαία στην Ευρώπη οι κοινέ ε, προτεραιότητες έχουν ε, τον τίτλο «Νέοι στην Ευρώπη». Τι μας αναμένει. Θα διοργανωθεί τον Απρίλιο στη Σόφια ένα συνέδριο με το θέμα αυτό ε, οι προκλήσεις ενώπιον των οποίων ε, βρίσκονται οι νέοι, καθώς και η συμπερίληψη της, ε, των δικών τους προσδιοκιών για τη χάραξη της προσεχούς ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους νέους. Χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση των στοιχείων κλειδί στο, στην πολιτική για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα τις πολιτικές προτεραιότητες και να ξεπεράσουμε τις, τα, τις προκλήσεις για τους νέους σημαντικά προβλήματα το πλαίσιο Ευρωπαϊκή Συνεργασία, η, το 17-18 η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία είναι το πιο σημαντικό πολιτικό εργαλείο για τους νέους. Θα εξετάσουμε λοιπόν το πλαίσιο αυτό μέσω των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να χάξουμε μια νέα στρατηγική στο πρώτο ήμιση του έτους 2018. Η Βουλγαρική Προεδρία οργανώνει συζητήσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες ε, μέλη να επεξερθούν στις δικές συστάσεις για τη στρατηγική αυτή και να τις υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα θέμα κλειδί είναι και ο φάκελο για την ε, Ευρωπαϊκή Ελληνική. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να συντείνει στην πρόθεση των ευρωπαϊκών αξιών καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών διεξιοτήτων στους νέους ανθρώπους. Όλα αυτά μπορούν να περάσουν θετικά την προθυμία τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να επηρεάσει και τις δυνατότητες απασχόλησης. Ε, το Δεκέμβριο του 2017 το Συμβούλιο έλαβε την εντολή για διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Η Βουλγαρική Προεδρία είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τι ολοκληρώσει. Αναμένουμε την ανάθεση εντολή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Εκτιμούμε ιδιαίτερω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση και ανάληψη πρωτοβουλειών για την αποτελεσματική εξέλιξη της πολιτικής των νέων και της συμμετοχής της νεολαίας. Έχουμε μια προβλέψιμη πολιτική συζήτηση σε υψηλότατο επίπεδο για το, με θέμα το ρόλο των νέων ανθρώπων για την εφαρμογή των στόχων για, την βιώσιμη, ε, για τους βιώσιμους στόχους των Ηνωμένων ε, Εθνών. Ε, στον τομέα του αθλητισμού, εδώ η έμφαση δίνεται στην πρόθεση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού. Το μέλλον Ευρώπης και, της Ευρώπης και των αξιών της έχουν ζητηθεί σε υψηλότερο επίπεδο. Αλλά και σε ε, άτυπο επίπεδο το Σεπτέμβριο του 2017 στην Πρατισλάβα, το 2016, συγγνώμη, ο καθώς και την ε, συνάντηση των επικεφαλής κυβερνήσεων στη Ρώμη με ευκαιρία της 20 υποπετίου υπογραφής των συνθήκων της Ρώμης. Το σημαντικότερο μήνυμα που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι η πρόσβαση των αθλητισμό συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων γιατί ενισχύει τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στον αγώνα κατά τη ριζοσπαστικοποίηση και τη αποφυγή τη επιθετικότητας. Η Βουλγαρική Προεδρία θα θέλει να επεξεργαστεί μια απόφαση του Συμβουλίου στον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί στην ε, συνάντηση του Συμβουλίου το Μάιο του 2018. Σημαντικό εδώ είναι το θέμα του μαζικού αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής ε, ένταξης ε, και θέλουμε να δείξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς ε, παραδοσιακά αθλήματα μπορούν να βρουν τη θέση τους και στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και να είναι και φορείς παραδοσιακών αξιών. Η Βουλγαρική Προεδρία θα εξετάσει το θέμα της χειραγώγησης του της, ε, της νόθευσης των ε, αποτελεσμάτων στον ε, αθλητισμό, των επιδόσεων και του ντόπινγκ. τα, τους επόμενους έξι μήνες θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Στις 24 και 25 στη Σόφια έχει διοργανωθεί ένα σεμινάριο με θέμα την αποφυγή του ντόπινγκ στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων και την άμβληση του φερμένου αυτού μέσω της εκπαίδευσης. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι καλύτερη, το καλύτερο εργαλείο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ για επαγγελματίε όσο και για τεχνές είναι ε, ο, ο, μια εξαρτία διαφωτισμού. Χρειαζόμαστε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα αντι-doping για τους αθλητές, για τους ε, προπονητές, τους γονείς, αλλά και τους ερασιτέχνες αθλητές και τους πολίτες. Μία νέα μέθοδος στην πρόληψη του ντόπινγκ, η οποία θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω, είναι οι έρευνες που γίνονται ε, για την ε, ανείχνευση του ντόπινγκ συνδέοντας ρυθμιστικά, ρυθμιστικές ε, διατάξεις με την απαγόρευση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων. Ε, το μέλλον ενός διεθνούς συστήματος αντιτόπικ ε, βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει εδώ να συμβάλλει στη συζήτηση αυτή μέσω ενός σωστού συντονισμού και μιας καλής παρουσίας των κοινών προβλημάτων στην ε, συνεδρίαση της Παγκόσμιας ε, Οργάνωσης για το αντι Η παγκόσμια αυτή οργάνωση έχει, ολοκληρώ... έχει ξεκινήσει την πρώτη φάση εκπόνησης ενός νέου ε, δεοντολογικού κώδικα και η Βουλγαρική Προεδρία αναμένει την... Ε, θα επεξερθεί συγγνώμη, την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είμαι περήφανος που η Βουλγαρία στο πρώτο ημίση του 2018 θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπόνησης μιας κοινή ε, στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκπόνηση του κώδικα αντι-doping. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι στην εργασία μας στον τομέα του αθλητισμού και της νεολαίας θα εργαστούμε σύμφωνα με την αρχή να λάβουμε υπόψη μας τα επιχειρήματα όλων των ενεχόμενων ούτως ώστε να πετύχουμε ε, αποτελέσματα για όλους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κράλεφ και τώρα θα έρθουμε ε, στην Υφυπουργό κυρία Γκρέσεβα που έχει το λόγο για 15 λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Εκπαίδευσης, ε, είναι τιμή μου ε, που πάρθαμε εδώ επ' ευκαιρία της ανάληψης Βουλγαρικής Προεδρίας για να παρουσιάσω το πρόγραμμά μας για τους επόμενους έξι μήνες στον τομέα του πολιτισμού. Δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε επισκεφθεί τη χώρα μας, αλλά η χώρα μου, η χώρα μου έχει μια χιλιετή ιστορία. Ε, συγκαταλέγεται στις, ε, στα πιο παλιά ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό το οποίο έχει εδραιωθεί είναι η πεποίθηση ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι διαφορές και η πολιτιστική ποικιλομορφία συνιστά ύψιστη αρχή την οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε και να μεταβάσουμε στις επόμενες γενναίες. Η Βουλγαρία αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια πολύ σημαντική συγκυρία. Σήμερα το ευρωπαϊκό εγχείρημα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ υψηλό βαθμό συνοχής, κοινέ αξίες και μια καινούρια φρέσκια ματιά στο μέλλον. Για μας ο πολιτισμός ε, είναι ένα από τα δοκιμασμένα εργαλεία που οδηγούν στην ανάπτυξη, ε, στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, η οποία ε, είναι συνιστά κάτι περισσότερο από μια κοινή αγορά στην Ευρώπη. Γι' αυτό ο πολιτισμός κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή βασίζεται σε μια ε, νέα αντίληψη όσον αφορά την κοινή μας ευρωπαϊκή ιστορία. Οι προτεραιότητες θα δοθούν στους πολίτες, στους νέους ανθρώπους... τη δημιουργικότητα και το δυναμικό ψηφιοποίηση. Η Βουλγαρική Προεδρία διατύπωσε τέσσερις προτεραιότητες... για το, το μέλλον της Ευρώπης και των νέων ανθρώπων, ε, κοινωνική προσέγγιση, ανάπτυξη ευημερία. Ε, ε, συνοχή των Δυτικών Βαλκανίων και ασφάλεια σε μια Ενωμένη Ευρώπη, ε, ψηφιακή οικονομία, η συνεργασία μας στο χώρο των οπτικοκοστικών βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με αυτές τις προτεραιότητες και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη και στην τελευταία προτεραιότητα η εξέταση της οδηγίας για τα, τις οπτικοστικές υπηρεσίες συνιστά προτεραιότητα της ε, Προεδρίας μας. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία αυτής της οδηγίας και τη βαρύτητα μιας ε, γρήγορης ε, εξέλιξης για την εύρυθμη λειτουργία μιας ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής ε, αγοράς. Επιτρέψατε μου να πω ότι κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής, της Μαλτεζικής και της Εστανικής Προεδρίας ε, πήκαν ε, οι προϋποθέσεις ε, για την πρόοδο εδώ και θα ήθελα να τις ευχαριστήσω ιδιαίτερα και αυτή τη στιγμή το ίμιση των άρθρων της οδηγίας έχει εξεταστεί σε πολλά σημεία, έχει επιτευχθεί μια συμφωνία. Μεταξύ αυτών των άρθρων συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, οι διατάξεις για μια βελτιωμένη πρόσβαση στα οπτικοακουστικά περιεχόμενα για άτομα με αναπηρίες, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αυτονομίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στον οπτικοακουστικό τομέα, η διατάξη της Ευρωπαϊκής ε, Ομάδας για τη ρύθμιση του οπτικοακουστικού τομέα που θα φροντίσει για μια καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας και οι διατάξεις για τη δημιουργία μιας ε, κοινή ε, τράπεζας οπτικοακουστικών δεδομένων. Η Προεδρία μας θα ε, θα επικεντρωθεί στις προσπάθειές της ε, για αυτό το σημαντικό νομοθέτημα και το ίδιο ισχύει και για τις ε, διατάξεις που αφορούν την καλή λειτουργία της ε, αρχής της, ε, του κράτους ε, προέλευσης καθώς και της προστασίας των οπτικοακουστικών περιεχομένων. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πετύχουμε μια συμφωνία για τις διατάξεις αυτές. Επίκυνται βεβαίως συζητήσει για δύο σημαντικά θέματα. Η πλατφόρμα για τα περιεχόμενα των βίντεο ταινιών πολύ σημαντικό θέμα προκειμένου να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικό συμβιβασμός. Έχουν γίνει οι πρώτες τεχνικές επαφές ε, αρχές Ιανουαρίου και ήταν αισιόδοξε οι προοπτικές. Επιτρέψατε μου ε, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες γιατί η εξέταση της οδηγίας δεν είναι εύκολο έργο. Παρ' όλα αυτά είμαι πεπισμένη ότι στο πνεύμα της ε, σωστής συνεργασίας και της εμπιστοσύνης θα μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία για το φάκελο αυτό, για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας. Για μας είναι σαφές ότι τόσο η ποιότητα όσο και ο ρυθμός είναι εξίσου σημαντικά θέματα. Θα προσπαθήσουμε να τα πετύχουμε στο πλαίσιο μιας καλής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε πεπισμένοι ότι από κοινού μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό προκειμένου να έχουμε ένα νομοθέτημα το οποίο θα είναι χρήσιμο ε, στους ε, καταναλωτές και τους δημιουργούς ε, μιας κοινή ευρωπαϊκής κληρονομιάς προκειμένου επίσης να προστατευθούν και τα δικαιώματα των δημιουργών. Μια άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι το, η πολιτιστική κληρονομιά όπως είπαμε. Για μας αυτό θα είναι ένα οριζόντιο θέμα και επιτρέψατε μου να σας ε, ευχαριστήσω για τις ε, προσπάθειες που έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες μέλη συνέβαλαν ενεργά στην ε, εξέλιξη και εφαρμογή αυτής της ιδέας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω προς τη δική σας Επιτροπή και την εισηγήτρια την κυρία Κώστα. Η πολιτιστική κληρονομιά χτίζει γέφυρες όχι μόνο στο, προς το παρελθόν μας, αλλά αφορά, είναι και ένας στρατηγικός πόρος για την, μια καλύτερη κοινωνική πραγματικότητα και μια βιώσιμη πολιτιστική εξέλιξη της Ευρώπης. Θα πρέπει να ζητήσουμε μια απάντηση στο ερώτημα τι ακριβώς σημαίνει η πολιτιστική κληρονομιά για τις κοινωνίες μας και για το μέλλον της Ευρώπης από τη μία θα εξετάσουμε το ρόλο της πολιτικής κληρονομιάς όσον αφορά την επίτευξη στόχων των άλλων ε, πολιτικών της Ευρώπης και της κοινωνίας. Θα αναστήσουμε μια απάντηση στο ερώτημα πώς θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις επιμέρους πολιτικές της ε, πολιτικής κληρονομιάς και να τις ε, εξισώσουμε ε, Θέλουμε στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες ε, πολιτικές. Ε, το Μάιο του 2018 θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σε επίπεδο κορυφής. Ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης κάποια περιεχόμενα τα οποία θα διαφυλεχθούν ως πολιτιστική κληρονομιά για τις επόμενες γενναίες. Αυτό θα είναι ένα από τα θέματα στις, το Μάιο γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε τους υπουργού μια συζήτηση για, την, ε, για το μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ε, πολιτιστική κληρονομιά. Από όλες τις χώρες υπάρχει υποστήριξη για την πολιτιστική κληρονομιά. Από εκείνες τις χώρες που επέγραψαν την ε, Συμφωνία του Νταβός. Σε λίγους μήνες θα παρουσιαστεί το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, εντός το οποίο ορίζονται προτεραιότητες για τα επόμενα έξι χρόνια. Επιθυμούμε να συμπεριληφθεί εδώ και ο πολιτισμός, γιατί λειτουργεί υπέρ της συνοχής της ευρωπαϊκής κοινωνίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ε, ποικιλομορφίας καθώς και της δημοκρατίας. η σημασία του πολιτισμού για το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι καθοριστική και αυτό τόνισε και το Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο. Ε, αφετηρία για τη χρηματοδότηση των πολιτιστικών προγραμμάτων θα είναι η διάμεση αξιολόγηση και με αυτήν συνδέεται η επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Προγράμματος που υπάρχει εδώ και δέκα χρόνια. Σε μια συγκυρία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις, ο πολιτισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ζωογονεί τις πόλεις και τις περιφέρειες, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ε, λειτουργεί σαν έμβλημα για πετυχημένες και δημιουργικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναζωογονήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα, γιατί ο πολιτισμός ισοδυναμεί με έμπνευση που τόσο χρειαζόμαστε, χτίζει γέφυρες μεταξύ των γενναιών. Ένα από αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα που αποτελείται από μουσικός από όλες τις χώρες ε, μέλη. Η Κομισιόν ε, υπέβαλε μία ε, σχετική πρόταση για χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Τον τελευταίο Δεκέμβριο οι χώρες έλαβαν το η, εντολή, η την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα όσον αφορά ε, την, το έργο της και ελπίζω να υπάρξει σύντομα μια συμφωνία μεταξύ μας. Τον Ιούνιο του 2016 είπα ότι εκπρόσωπος από κοινού με την Επιτροπή πρότεινε μια προσέγγιση η οποία θα βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για διεθνείς σχέσεις στον τομέα του πολιτισμού. Στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού το 2015 βεβαίωσε ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Συμβούλιο ε, αποφάσισε τη δημιουργία μιας ε, πλατφόρμας για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στον τομέα του πολιτισμού. και ξεκίνησαν σχετικέ δραστηριότητε τον περασμένο Ιούνιο. Η Βουλγαρική Προεδρία πρόκειται να στηριχθεί στην εργασία των προηγουμένων Προεδριών και να τι οριστικοποιήσει. Αφού η αρχική εντολή λύγει τον Ιούλιο αυτού του έτους, θα πρέπει να συζητήσουμε τις χώρες μέλη ε, και την Επιτροπή για την επεξεργασία μιας ε, σταδιακής ε, προσέγγισης όσον αφορά της διεθνούς ε, προσέγγισης στο χώρο του πολιτισμού. Όλα τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν στις διεθνείς διοργανώσεις στο πλαίσιο της ε, Προεδρίας μας. Το Φεβρουάριο θα έχουμε μια άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα ο πολιτισμός σαν ε, σφαιρική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης θα έχουμε μια συνάντηση με τις χώρες Άζιαν που θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική κληρονομιά σε σχέση με τις επιχειρήσεις κλπ. Επίσης ε, τα τέλη, στα τέλη Μαρτίου στο Plovdiv θα υπάρξει ένα συμπόσιο. Το Plovdiv είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2018 και θα χαιρόμουν να σας ε, καλωσορίσω στη Βουλγαρία. Ένα άλλο θέμα είναι το δικαίωμα των, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, προβλέπονται δύο νομοθετήματα για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των δημιουργών Θα στηριχθούμε στην, στο έργο της προηγούμενης Προεδρίας εδώ, η οποία σημείωσε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την επιτεύξη συμφωνία στο Συμβούλιο. Στις 15 Δεκεμβρίου επιβάθηκε εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τα πνευματικά δικαιώματα, όσον αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Ε, αυτή τη στιγμή τρέχουν οι διοργανικές, ε, επόμενο μήνα συγγνώμη, θα ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να υπάρξει πολιτική συμφωνία για το σημαντικό αυτό ντοσιέ γιατί ε, το, η έμφαση θα δοθεί σε δύο σημαντικά ερωτήματα. Η εισαγωγή ενός δικαιώματος για τους δημιουργούς και για τις ε, υπηρεσίες των, ε, της κοινωνίας, ε, στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορικής. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τις διαφορετικές ε, ευαισθησίες των διαφόρων ε, ενεχόμενων ε, δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί συνένεση. Μόνο εφόσον το Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφωνήσουν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διοργανικές διαπραγματεύσεις που μάλλον θα γίνει στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 ε, και πάλι θα ήθελα να εκφράσω την, ε, την ε, επιθυμία μου για μια καρποφόρα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα χαρώ πάρα πολύ, όπως είπα, να σας δω στη χώρα μας, στο εναρκτήριο Γκαλά της Βουλγαρικής Προεδρίας την 1η Φεβρουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες, σας περιμένω βεβαίως. Και επίσης τα εγγένεια της έκθεσης για δημιουργικά προγράμματα και επικοινωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κράλεφ και κυρία Κρέσεβα. Τώρα θα περάσουμε στο γύρο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις. Είπατε εν συντομία πόσο σημαντικό είναι το έτος της προσπάθειας αυτές. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια συνείδηση για την ευρωπαϊκή πολιτική κληρονομιά. Δεύτερον, αναφερθήκατε στο μεσοπρόθεσμο δημοσιο... Δεν, μπήκαν, δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ε, στον ε, ε, και σας άποψη εδώ. Ευχαριστώ, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για ακρόαση το απόγευμα, γιατί θέλουμε να δώσουμε στρατηγική σημασία για την πολιτική για την νεολαία, όχι μόνο στα προγράμματα ε, και όχι μόνο κάθετα, αλλά και πιο οριζόντια. Ε, βασιζόμαστε λοιπόν στην Βουλγαρία για μια πιο καλή προσέγγιση. Τώρα, ο αθλητισμός ελπίζουμε να προωθήσετε στη διάρκεια της Προεδρίας σας την φορά την πραγματικότητα του αθλητισμού και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς ε, θέλετε να κάνετε από πλευρά Συμβουλίου εθελοντισμός και αλληλεγγύη. Εμείς εργαζόμαστε εντατικά. Εγώ είμαι συγγήτρια για το Ευρωπαϊκό Σώμα ή Υπηρεσία Αλληλεγγύης ε, και θέλουμε να έχουμε μία βάση εθελοντισμού γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένη. Καταρχάς, αύριο θα γίνει ο τριμερής διάλογος ε, και ελπίζουμε να μπορούσουμε να έχουμε μια καλή συμφωνία. Τώρα, για το VMS, για μας είναι πάρα πολύ σημαντική να εγκριθεί η οδηγία για το ακουστικά μέσα, γιατί εμείς ελπίζουμε και σε αυτή την οδηγία και στην ε, διαδικτυακών ε, μέσων, τις πλατφόρμες δηλαδή που υπάρχουν για το περιεχόμενο και των δικαιωμάτων των δημιουργών να είναι σε ισορροπία και να δοθεί ιδέουσα προσοχή. Ελπίζουμε λοιπόν και στη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας και με τον Επίτροπο να υπάρχει καλύτερη σχέση μεταξύ ε, ψηφιακών θεμάτων πολιτισμού νομιάς. Ξέρω ότι ε, δεν υπήρξε επαρκής δέσμησης. Υπάρχει το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση της πολιτικής ε, κληρονομιάς και κοινέ αξίες δεν με 0,2% ε, του προπολογισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό, είναι πολύ χαμηλό. Διάβασα ένα άρθρο του βουλγάρου ε, φιλοσόφου Κάστευστο Σπίγκελ αυτή την εβδομάδα που είπε ότι θα πρέπει να είναι λόγος να νιώθουν ανώτεροι. Ε, καλωσορίζω αυτή την προσέγγιση γιατί νομίζω ότι αποκαλεί πολύ καλό σημείο για να υπάρχει κοινή συνονέωση στην Ευρώπη μεταξύ Δύσης και Ανατολής ε, και της λεγόμενης ε, ε, ισχύς, ε, ισχυρής χώρας της Ευρώπης, της χώρας μου της Γερμανίας. Ε, για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είπα ήδη ότι θα ήθελα να λέγεται Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αλληλεγγύης γιατί υπήρχαν κράτη-μέλη που δεν ε, ε, ήταν σύμφωνα με τον όρο σώμα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, ιδίω για του νέου ανθρώπου, για να υπάρχει αλληλεγγύη και με τι προσεχεί εκλογέ ε, το 2019 ελπίζουμε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και να του πείσουμε να ψηφίσουν. Και κάτι τελευταίο. Η μεταρρύθμιση για τα πνευματικά δικαιώματα. Η Επίτροπο ε, Μαρίσα Γκαμπριέλ ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό όπω και, και εγώ και να σα πω ότι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να καταλάβουν οι Αμερικανοί ότι οι ψηφιακέ πλατφόρμε πρέπει να φορολογούνται, επομένω πρέπει να πληρώνουν φόρους ε, και κατά την άποψή μου χρειάζεται ένας ψηφιακός φόρος. Χρειάζεται μια υποχρέωση αδειοδότησης, όσο, όχι τόσο όσο προς τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά υποχρέωση αδειοδότησης και να αναφέρεται αυτό στο άρθρο 9, ώστε η εμπορική χρήση, αν δεν έχει δημιουργηθεί το περιεχόμενο από την πλατφόρμα, να υποχρεούνται να ε, πληρώνουν φόρο και να υπάρχει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, Επίσης, πλατφόρμες οι οποίες ε, ε, προσδίδουν τίμημα σε πολιτιστικό περιεχόμενο θα πρέπει να κάνουν συμφωνίες αδειοδότησης με οργανισμούς οι οποίοι ε, μεταρρυθμίστηκαν από πλευράς μας και πρέπει να έχουν και ευθύνε για τα fake news, τις ψευδείς ειδήσει και ε, τη ρητορία μίσους. Αν υπάρχει κοινή προσέγγιση στο Κοινοβούλιο, μπορούμε να δείξουμε και στους ψηφοφόρους ότι ε, μπορούμε να κάνουμε κανές κινήσεις και έξυπνη νομοθεσία προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα έχουμε, θα ακούσουμε τις ε, υπόλοιπες παρεμβάσεις. Παρακρότω, ο Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγώνων ε, για την επικύρωση της σύμβασης του Μάκολεν και τη χειραγώγηση αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά ατυχές. Έχω την εντύπωση ότι τελικά θα χαθεί αυτή η ευνοϊκή συγκυρία για να υπογράψουμε και να επικυρώσουμε αυτή τη σύμβαση, ενώ το πρόβλημα των στημένων αγώνων προωθεί τις, ε, την κοινή, τις κοινές αξίες μας στον αθλητισμό η παρούσα κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ξενοφοβία, η ζωσπαστικοποίηση, η δημοσιολαβητή σκοπεύεται ε, να διευκολύνεται, ε, να επιληθεί το πρόβλημα που και της ΦΥΜΠΑ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκο. Με το σημαντικό αυτό ντοσιέ για τους ε, νέους, το που αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Γιατί στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Σημαντική υστέρηση. Ευχαριστώ. Κράλεφ. Αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχετε συνείδηση ότι εδώ δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα για την νεολαία που είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, δεν προβλέπονται να φεμάξουμε το Εράσμους. Θέλουμε ένα, μια καινούρια χρηματοδότηση, άλλα κονδύλια. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε αυτό το θέμα και να παλέψετε για την αύξηση των κονδυλίων, ούτως ώστε το Εράσμος να παραμείνει σταθερό για την εκπαίδευση των νέων ε, χρηματοδότησης. Ο προκάτοχος στο Συμβούλιο δεν μπόρεσε να το πετύχει. Το Συμβούλιο Υπουργών μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δεν αύξησε τα, τους πόρους. Μία Αντίστοιχη έκκληση ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Έτο ε, Κοινή Πολιτιστική Κληρονομιά. Θέλουμε να πολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Είναι οι κοινέ μα πολιτιστικέ ε, αξίε, η πολιτιστική μα κληρονομιά. Αυτό είναι ο στόχο αυτού του έτου. Και θα ήθελα να σα ε, παρακαλέσω να εξετάσετε πώ μπορείτε να αυξήσετε το προπολογισμό. 8 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προπολογισμό και να αξιοποιηθούν ιδιαίτερω για τους νέους. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγα λεπτά χρόνο για τις απαντήσεις και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αντίστροφη σειρά με την κυρία Υφυπουργό. Παρακαλώ έχετε το λόγο ε, ή δυνατόν να είστε αρκετά, να συμπυκνώσετε τα λεγόμενά σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις και επειδή πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να συνοψίσω τα ερωτήματα αυτά στις απαντήσεις μου. Η πολιτιστική μας κληρονομιά, η διατήρησή της, τα κονδύλια για την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να αυξηθούν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό αλλά και στους εθνικούς προπολογισμούς η Κομισιόν πιστεύω θα το λάβει υπόψη της. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πολιτιστική κληρονομιά να θεωρηθεί ε, κοινή υποδομή, να μπορέσουν ενισχυμένα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της ψηφιοποίησης και να έχουν το αίσθημα ότι ανήκουν ε, στην Ευρώπη αλλά και στις δικές τους χώρες. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έτους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς στη Βουλγαρία, μόνο τους πρώτους τρεις μήνες. Για μένα θα ήταν σημαντικό να ενισχύσουμε περισσότερο τις Ευρωπαϊκές ημέρες της πολιτιστικής κληρονομιάς και αυτό συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά γεγονότα ε, για την πολιτιστική πολιτιστικής πρωτεύουσας. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, σημαντικό είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στην, θα αναφερθεί στην έκθεση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος ε, Δημιουργική Ευρώπη. Έχουμε περισσότερα, προγραμματίσουμε περισσότερα κονδύλια για την επόμενη περίοδο. Ελπίζουμε επίσης ότι θα έχουμε μια φιλόδοξη προσέγγιση για την περίοδο μέχρι το 2020 και να... Όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Τρίπελ για τα πνευματικά δικαιώματα, θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές καθώς και για τους ε, πολιτιστικούς δημιουργούς, ιδιαίτερο στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και εσείς για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βουλγαρική Προεδρία πρόκειται να επεξεργαστεί περαιτέρω το θέμα αυτό του copyright και αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα δημιουργικά περιεχόμενα και θα εκπονήσουμε και κάποιους ε, κανόνες για τους φορείς τέτοιων περιεχομένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κράλεφ, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο και τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερως ενδιαφέροντα. Οι ερωτήσεις που έλαβα είναι πολύ ενδιαφέρουσες που θα συμβάλλει στην πρόθεση των ευρωπαϊκών αξιών και των ικανοτήτων των νέων ανθρώπων. Μόνον έτσι μπορούν οι νέοι άνθρωποι να μπουν στην αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο συζήτησε την πρόταση της Επιτροπής και θέλουμε στο πλαίσιο της Προεδρίας μας να καταλήξουμε σε μία ενιαία τοποθέτηση. και τη δυνατότητα εθελοντικής εργασίας των νέων ανθρώπων, θα ήθελα να πω ότι το υποστηρίζουμε αυτό πλήρως. Το θέμα ε, στρατηγική για τους νέους είναι μια περιττέρω προτεραιότητα για μας. Για την Προεδρία είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό το ονομένο πλαίσιο να μπορεί να στηριχθεί σε μια στρατηγική. Μόνον έτσι μπορούμε να προωθήσουμε μια βιώσιμη πολιτική στον τομέα της, ε, των νέων, της νεολαίας. Οι καταλεκτικές ε, ε, τα, τα συμπεράσματα μάλλον του Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική της νέας οι καταλεκτικές τα, τα συμπεράσματα μάλλον του Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική της 2018 πρόκειται να διοργανώσουμε ένα συνέδριο για, ως ε, πλατφόρμα και δυνατότητα για τους νέους προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι συστάσεις αυτές πρόκειται να συμπεριληφθούν στη νέα στατική για την νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο κ. Μποκτανπρίν έθεσε το ερώτημα αυτό εν σχέση με την χειραγώγηση των αθλητικών αποτελεσμάτων. Το θέμα αυτό βεβαίως έχει μια, διεθνή, έχει μια βαρύτητα διεθνώς. Είναι σημαντικό πρόβλημα για πολλές χώρες. Γι' αυτό ε, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης οργανώσεις που αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών ε, αποτελεσμάτων όπως οι υπηρεσίες της Ιντερπόλ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε προγραμματίσει μια συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων με τίτλο ε, «Καιρεότητα», συνεδριάζει στη Βάρνα και έχει σε στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την διεθνή συνεργασία στο επίπεδο της πρόληψης, της χειραγώγησης στον αθλητισμό. Πρόκειται να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά την ε, χειραγώγηση των ποδοσφορικών αγώνων Και έχει υπάρξει μια συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014. Η Βουλγαρική Προεδρία θα εξετάσει τις νέες προτάσεις και το πώς μπορούν να, να ε, διαμορφωθούν από το Συμβούλιο. Αυτό θα είναι σημαντικό βήμα για την πρόληψη χειραγώγηση των αθλητικών αποτελεσμάτων. Европейската лига. Разбира се, това е много тежък въпрос, който може да засегне не само. Όσον αφορά τη ФИБА, έχουμε οργανώσει κάποιε συναντήσει με εκπροσώπου τη. Η βουλκαρική πλευρά δεν έχει έτοιμη μία λύση, αλλά μπορούμε να λειτουργήσουμε ως διαμεσολαβητές. θα Η Βουλγαρική Προεδρία έχει την άποψη ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να συμβάλλει ε, και την, ε, τη μυσαλλοδοξία και την ξενοφοβία. Θα υπάρξουν κάποια από τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, αλήθεια, είναι πολύ ε, λίγος ο χρόνος. Γιατί στην Επιτροπή μας έχουμε ένα ευρύ φάσμα ποικίλων θεμάτων. Γι' αυτό ποτέ δεν μας φτάνει ο χρόνος αλλά πραγματικά επενδύω σε μια αποτελεσματική και επικοδηματική συνεργασία της Επιτροπής με τη Βουλγαρική Προεδρία και εγώ ελπίζω πάρα πολύ να έχουμε την υποστήριξη της Βουλγαρικής Προεδρίας για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την διαμόρφωση των μελλοντικών προγραμμάτων συμπεριλαμβανόμενου και του Ευρωπαϊκού Σώματος ε, Ελεγγύης. ούτω ώστε εδώ να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο προκειμένου να γίνουν επενδύσεις και να αυξηθούν μάλλον οι επενδύσεις για τους νέους για να αυξηθεί και η συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά επενδύουμε σε μια... στην υποστήριξή σας. Σε ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Καλημέρα σας.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 Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συνεδρίαση, οπότε σας παρακαλώ όσοι βγαίνουν από την αίθουσα να το κάνουν αυτό γρήγορα και ήσυχα. Φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της μέρης διάταξης ε, για το πρωί τουλάχιστον και εδώ τώρα θα μιλήσουμε για τα σχέδια υποστήριξης ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης που σχετίζονται με την ε, γίνεται η ε, προσκεκλημένη μας. Hello. Hello.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 Έχουμε δύο project που θα μας παρουσιάσουν σήμερα, μας παρουσιαστούν σήμερα. Ε, ο στόχος είναι να... Λοιπόν. Έχουμε δύο project που θα μας παρουσιάσουν σήμερα, μας παρουσιαστούν σήμερα. Ε, ο στόχος είναι να προωθήσουμε τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ε, για ευρωπαϊκά ζητήματα. Ξέρουμε ότι η ελευθερία του τύπου, ο πλουραλισμός... Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να μεταδίδουμε ειδήσει και μάλιστα αξιόπιστες ειδήσει για ευρωπαϊκά ζητήματα. Ε, θα... Οι προκλήσεις είναι πολλές. Μόνο από κοινού μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η οποία είναι project manager, για το Ευρωπαϊκό News Hub Ευρωπαϊκών Δεδομένων από την Ακάρντο ο οποίος είναι πρόεδρος του Fox Ευρώπη. Λοιπόν, Μάρτιν Ντόσεν πρώτα για μέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κατέστη εφικτό δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν νιώθουν ότι ενημερώνονται επαρκώς για ευρωπαϊκά ζητήματα. Από την άλλη, πολιτές στο δημοσιονομικό πρόγραμμα υπήρχε μεγάλη ανάγκη, ε, μεγάλη ζήτηση ενημέρωσης ε, για ευρωπαϊκά ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως ε, τα χρήματα που είχαν διατεθεί για τη χρηματοδότηση δηλαδή μέσων επιγραμμικά, εκεί όπου όλο και πιο συχνά βρίσκονται οι αναγνώστες, ιδιαίτερα η νέα γενιά, τα γεγονότα σε μια εποχή ψευδών ειδήσεων. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η ποιότητα, να βελτιωθεί η ποιότητα της, δημοσιογραφία και να έχει πρόσβαση σε όρια. Οι συνάδελφοι από τα πρακτορία ειδήσεων μας είπαν πάλι σήμερα το πρωί ότι χρησιμοποιούν από κοινού τους πόρους έτσι αυξάνεται η δυνατότητα κάλυψης ειδήσεων υπάρχει το ε, new δηλαδή ε, σε επίπεδο μέσων ενημέρωση στην Ευρώπη στο σύνολό του. Και βεβαίω το θέμα είναι να φτάσουμε στον πολίτη, να βελτιώσουμε την ποιότητα της συζήτησης και της ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτά είχα να πω εγώ. Νομίζω ότι μπορεί να μιλήσουν και οι επόμενοι ομιλητές από εδώ και από την ΤΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση του, Ευρω... του, του News Hub μάλλον ε, των Ευρωπαϊκών Δεδομένων με την ANSA σελίδα με δεδομένα ε, για ευρωπαϊκά ζητήματα και σχετικές ειδήσει. Ε, πρόκειται για το News Hub ευρωπαϊκών δραστικά γραφικά, γραφήματα προσπαθούμε να προωθήσουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα που συζητώνται σε ευρωπαϊκό μέσο των πρακτορείων ειδήσεων προς όλα τα μίντια. Όλα τα στοιχεία αυτά μπορούν να δημοσιευθούν, ώστε να μπορούν οι αναγνώστες να καταλάβουν πιο εύκολα δύσκολα δεδομένα. Ε, μπορούμε να προωθήσουμε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Ε, πρόκειται για φόρμα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο εύκολα ε, διαδραστικά και στο διαδίκτυο. Όλα αυτά, αυτό ε, είναι πραγματικά, πραγματικό περιεχόμενο πολυμέσων, το οποίο είναι φιλικό προς το διαδίκτυο. Έχουμε διάφορες τεχνικές δεδομένων ε, και αυτό προσθέτει προσθέμενη αξία στις πληροφορίες που δίνουμε. Θέλουμε να έχουμε τις φορές από την εκδοτική ομάδα για τη μετανάστευση, για το Brexit, αλλά και για το θέμα της Ευρωζώνης. Οι πληροφορίες, ε, επίσης χρησιμοποιούμε ε, το πολύ ισχυρό δίκτυο Twitter που υπάρχει γενικότερα είναι πιο εύκολα κατανοητά από τους πολίτες. Το αποτέλεσμα θα είναι, ελπίζουμε, ότι το News Hub θα βοηθήσει για τη διαφάνεια, θα βοηθήσει ε, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό την ερχόμενη θητεία. Επίσης θα συνεχίσουμε την προσπάθεια marketing στέλνοντας πολλά, πολλά Επίσης θέλουμε να συνεχίσουμε την υποδομητική συνεργασία που ξεκινήσαμε μεταξύ των πρακτορείων των εθνικών, των εθνικών και να συναντιόμαστε πιο συχνά. Και... Ε, είναι η επόμενη μιλήτρια, όχι. Ωραία, η Κιέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα σας παρουσιάσω το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, δημοσιογραφίας δεδομένων, να περιμένουμε λίγο να ανοίξουν και οι διαφάνειες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο λοιπόν ε, ε, Δημοσιογραφίας Δεδομένων είναι μια συνεργατική πλατφόρμα για κάλυψη βάση δεδομένων των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Έχει ξεκινήσει από μια κοινοπραξία 16 πρακτορείων και υπηρεσιών από την Ευρώπη ε, από τον Νοέμβριο πέρσι ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας και ξεκινήσαμε με στόχο το συνδυασμό της παραγωγής των νέων και συνδυασμό των ε, μέσων που έχουμε, να έχουμε μια ενιαία φύγεται από τα δίκτυά μας και έχουμε και ε, πληροφορίες από τις πηγές για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και επικεντρωνόμαστε σε απλές δραστηριότητες ή συνεργασίες μεταξύ δημοσιογράφων. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα πάνελ για ε, συνεργατικές τέτοιες προσπάθειες. Προσπαθούμε να έχουμε μόνιμες σχέσεις και να βασιζόμαστε ε, σε αυτές τις συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων αιθουσών ε, τύπου και προσπαθούμε των δικτύων. Η παραγωγή ειδήσεων παρουσιάζει διάφορες μορφές, ε, οπτικοποίηση δεδομένων, βίντεο τα οποία θα ξεκινήσουν, ε, ερευνητική δημοσιογραφία μακροπρόθεσμα που θα ξεκινήσει, μπορούμε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πιο περίπλοκα δεδομένα και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα πρωτοτύπου περιεχομένου. Έχουμε και δημιουργία δεδομένων με πρόσβαση ε, σε ενδιαφέροντα αποθετήρια ε, δεδομένων ε, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα αυτά και να καλύψουμε ειδήσει και να υπάρχουν και καλές πρακτικές ανά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει και μία εικόνα ερευνητικής δημοσιογραφίας επεκτείουμε διάφορα θέματα και δεν εξετάζουμε τόσο το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Για παράδειγμα, υπήρχαν διάφορα... Επηρεάζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές η ίδια η κυρία Μέρκαλ και οι ιστορίες μας δημοσιεύονται και στην πλατφόρμα, αλλά αναρτώνται και σε πλατφόρμες ε, άρθρα τα οποία δημοσιεύσαμε. Έχουμε πάνω από χίλια, έχουμε διάφορες κάλυψη λόγω μετάφρασης και επαναδημοσίευσης. Τώρα, περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε δημοσιογράφους. Ένα από τα βασικά, για παράδειγμα, εργαλεία που έχουμε είναι το Stats Monitor, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που ε, αφορά data mining, εξόριση δεδομένων ε, και αυτή την εβδομάδα προσθέσαμε και μια ισπανική εκδοχή της ιστοσελίδας και τους επόμενους μήνες θα προσθέσουμε και άλλες γλώσσες μόλις ενταχθούν και νέα, νέα μέλη και θα τους παρουσιάσουμε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που παρουσιάζει το δίκτυο, για παράδειγμα ε, μεγάλες δημοσιογραφικές εκδηλώσεις ε, σας. Ε, εν τέλει, ούτως ή άλλως ο στόχος μας είναι το ευρύ κοινό να έχει περισσότερες ευρωπαϊκές ειδήσει ε, και ε, να υπάρχει μια συζήτηση βάση στοιχείων μέσω της δημοσιογραφίας για τα ευρωπαϊκά θέματα και να δώσουμε δυνατότητες σε δημοσιογράφους και να αυξήσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις ποιοτικές πληροφορίες. Ε, περικοπές για το Nets Plus, για παράδειγμα, δεν ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι εδώ στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Πολιτισμού και δημοσιογραφία βάση δεδομένων. Ε, αυτό το οποίο προκύπτει συχνά στην Επιτροπή μας είναι ε, το επίπεδο των ειδήσεων για την Ευρώπη. Ε, ε, άρθρα, για παράδειγμα, από κοινού να γίνεται μια συγκριτική μελέτη, διότι αν πραγματικά προσπαθούμε να πούμε ευρωπαϊκές ιστορίες και όχι μόνο ε, ευρωπαϊκά νέα με βάση την εθνική προοπτική. Σίλβια Κώστα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και το Κοινοβούλιο συνέβαλε για να βελτιώσουμε λίγο από τα, τα λάθη τα οποία έχουμε δηλαδή ε, στους δημοσιογράφους και χαίρομαι που η χώρα μου είναι εντός της πρωτοβουλίας με τη Λάνσα ε, να υπάρχει προσοχή για ευρωπαϊκά ζητήματα και να τεθεί και η Ευρώπη στο προσκήνιο όχι μόνο για αρνητικά θέματα. Είπατε ότι όλα αυτά είναι διαδραστικά. Πρόσβαση μέσω κωδικού. Ουσιαστικά υπάρχει δυνατότητα ελεύθερα να συμμετέχει κάπως ή πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες. Ε, και ενδιαφέρουν και το δίκτυο των δημοσιογράφων. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε επίσημες σχέσεις και έχετε υπάρξει ευαισθητοποίηση στο δημοσιογραφικό κλάδο στις διάφορες χώρες, γιατί πιστεύω ότι αυτοί μπορούν να αυξήσουν και αυτή την πρόσβαση, να μην είναι δηλαδή απλώς ατομική συμμετοχή, αλλά να συμμετέχουν και ενώσεις δημοσιογράφων ε, ε, επισήμως. Ευχαριστώ, η Χέλκα Ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε την προσέγγιση σας μαζί μας. Εχθές στη συνάντηση των συντονιστών μπορέσαμε να μιλήσουμε με εκπροσώπους ε, της Deutsche Welle και άλλους και φυσικά αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον διότι αναφέρθηκαν στο ίδιο ζήτημα πώς μπορούμε ε, να καταπολεμήσουμε τα fake news. Εγώ μίλησα και με τους εκπροσώπους της Google, τον ε, αντιπρόεδρο και τους ε, πρέσβεις ε, του Facebook ε, στο γραφείο μου το Δεκέμβριο και αναφέρθηκαν αυτές οι δυνατότητες αλγορίθμων για την καταπολέμηση των Facebook. Και το Google και το Facebook επέμεναν ότι δεν μπορεί να είναι μόνο τεχνική λύση, παρά το γεγονός ότι χρειάζεται το τεχνικό σκέλος, αλλά χρειάζεται και ο ανθρώπινος παράγων για να αποφασίσει τελικά μόνος του άνθρωπος τι είναι fake news και τι δεν είναι. Ε, το θέμα λοιπόν αυτό, ο συνδυασμός της ανθρώπινης ευθύνης και της ψηφιακής λύσης μέσω λογισμικού και αλγορίθμων, εάν φυσικά υπάρχει τέτοιο λογισμικό, ε, είναι το ερώτημά μου. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, γιατί το συζήτησα αυτό και με τον Φρεντερίκ Λεκλέρκ, ο οποίος είναι ο ε, αρχισυντάκτης ε, του EuroPTIF ε, μας είπε ότι μέχρι τώρα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις χρηματοδοτούν τη μάχη κατά των fake news και κατά την άποψή μου οι, οι ψηφιακές πλατφόρμες θα πρέπει να είναι υπεύθυνε και θα πρέπει να πληρώνουν αυτές και όχι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Εσείς τι πιστεύετε λοιπόν για τη χρηματοδότηση και ποια είναι η ευθύνη των ψηφιακών αμερικανικών μονοπωλίων, αν πρέπει να αναλάβουν και αυτοί κάποια ευθύνη. Και επίσης το όλο θέμα δεν είναι μόνο το μέλλον της ποιοτική δημοσιογραφίας στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι θα υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πληροφορίες οι οποίες ε, δεν θα ε, χρησιμοποιούνται με λανθασμένο τρόπο από εγκληματίες ε, και από τζιχαντιστές, για παράδειγμα, που εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά δίκτυα. Θα ήθελα να ξέρω πώς ορίζετε και πώς κάνετε διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων επιλογών. Ο κύριος Βέτα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των πολυμέσων και της χρηματοδότησής τους. Ε, ε, καλωσορίζουμε τις πρωτοβουλίες αυτές σε πολλές γλώσσες μάλιστα. Θέλουμε να αναπτύξουμε την δημόσια σφαίρα την ευρωπαϊκή. Θα ήταν καλό να επεκτείνουμε το πεδίο Τη δημοσιονομικής γραμμής για, τα, για τις δράσεις πολυμέσων, συμπεριλαμβάνοντας και πολιτιστικό περιεχόμενο. Παραδείγματο χάρη είναι υποτιτλισμός ε, πολιτιστικού περιεχομένου τηλεόρασης ανά την Ευρώπη. Αυτό έχει δείξει ότι ο υποτιτλισμός έχει πολύ θετικό ε, αποτέλεσμα στο να δημιουργείται ε, ευρωπαϊκό κοινό τηλεοπτικό. Μιλάμε για ποιοτικό υλικό και είναι πολύ φτηνός τρόπος πρόσβασης ε, σε πολιτιστικά αγαθά. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε ε, μια δράση follow-up για τον υποτιτλισμό του πολιτιστικού τηλεοπτικού περιεχομένου στα πλαίσια των δράσεων πολυμέσων και τη δημοσιονομική, γραμμή του 2019, διότι ε, θέλουμε να διαβρύνουμε όπως είπαμε, τη δημόσια σφαίρα, την ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. θα πρέπει να έχουμε ανεξάρτητες αξιόπιστες πληροφορίες. Το ερώτημά μου είναι ε, κατά πώς, τι, γίνεται μάλλον με τη μάχη κατά των fake news, διότι εάν θέλουμε να έχουμε πραγματικές, ε, ακριβείς πληροφορίες, αξιόπιστες, θα πρέπει να μπορεί κανείς να τις διαχωρίζει αυτές τις πληροφορίες από τις ψευδείς ειδήσει. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια εκστρατεία ολόκληρη κατά των fake news. Βραχυπρόθεσμα. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Έχετε κάποια στοιχεία για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά και πώς λαμβάνει η χώρα ε, και η ε, κατανομή, η γεωγραφική. Αφορά κάποιες χώρες ε, περισσότερο από άλλες θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται στη Τσεχία. Μάλλον αναφέρθηκε στον έλεγχο του περιεχομένου, του κατά πόσο δηλαδή οι ειδήσει είναι ψευδεί ή όχι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ε, με συγκεκριμένη προθεσμία ε, αρκούν, αρκεί αυτή η χρηματοδότηση ή αναζητείτε πηγές χρηματοδότησης και αλλού. Hub αφορά ένα ευρύτερο κοινό, δεν αφορά μόνο δημοσιογράφους αφορά το ευρύ κοινό. Για το δίκτυο δημοσιογράφων, το EDJ, αναφέρεστε πιο πολύ σε ένα πρόγραμμα δικτύωσης για τους δημοσιογράφους. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες από αυτόν. Έχουμε, μας μένουν 8 λεπτά, χωρίστε το χρόνο όπως νομίζετε εσείς καλύτερα και προσπαθήστε να απαντήσετε. Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το δίκτυο. Ναι, θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς ενδιαφέρει σε αυτό το δίκτυο. Ναι, θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς ενδιαφέρει σε αυτό το δίκτυο. Ε, Η IGNC είναι μια διεθνή, ένα διεθνές ζωγραφικό πρακτορείο. Έχουμε γραφεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γραφ... Ε, ασχολούμαστε με ειδήσει. Εργαζόμαστε καθημερινά ε, με βάση ε, την επικαιρότητα. τώρα όμως υπάρχει δυνατότητα να διαθέσει ένας, ένας διαθέσει χρόνο ένας δημοσιογράφος και να κάνει μια γενικότερη επισκόπηση του συμβαίνει στην Ευρώπη. Στο παρελθόν το γραφείο μας ε, στην Πολωνία έδειχνε, μας έλεγε ποια είναι η άποψη πολωνικής κυβέρνησης, ε, το γραφείο μας ε, στο Βερολίνο αυτό της γερμανικής. Τώρα όμως ε, υπάρχει δυνατότητα να εργαστεί κάποιος για μία εβδομάδα, για ένα φάκελο, με συνεισφορά από όλα τα γραφεία μας στην Ευρώπη, για να αναδειχθούν οι διαφορετικές απόψεις, για να μεταρρυθμίσει τη Ευρωζώνης, παραδείγματος χάρη, η δυσκολία του να υπάρξει σύγκληση ό,τι αφορά τη φορολόγηση, ε, για το θέμα της Google και της Amazon και το πώς μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Κάναμε ένα μεγάλο ρεπορτάζ γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πανέρχεται συχνά, αλλά είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από τους ε, πολίτες. Σε ό,τι αφορά αυτέ τι ε, έρευνε τώρα σε βάθο, το οποίο πανέρχεται συχνά, αλλά είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από τους ε, πολίτε. Σε ό,τι αφορά αυτέ τι ε, έρευνες τώρα σε βάθο, τώρα για τη συνεργασία μεταξύ πρακτορείων. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με την DPA, που ήταν ανταγωνιστή. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γαλλικά μιας και έχω το λόγο να το κάνω στις Βρυξέλλες ε, ε, που είναι πολύ και πιο σπάνιο για να απαντήσω στην κυρία Βεράιεν συγκριτικά με άλλα κράτη-μέλη και αυτό είναι εύκολο με βάση τα δεδομένα το data journalism είναι διαθέσιμα τα δεδομένα για να γίνει αυτή η σύγκριση επίσης φροντίζουμε πάντα ακόμα και αν προέρχεται ε, από έναν εταίρο μας το άρθρο που απευθύνεται φροντίζουμε πάντα ακόμα και αν προέρχεται ε, από έναν εταίρο μας το άρθρο που απευθύνεται